Good morning. No hammer. No hammer. Good morning. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι. Καλή σας μέρα επαναλαμβάνω. Κυρίες και κύριοι. Queridos colegas. Bonjour à tous. Good morning everybody and feliz año nuevo. Καλή χρονιά σε όλους, σε όλες τις γλώσσες. Good to have you back. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την πρώτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για το έτος 2013. Α ξεκινήσουμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στις 11 το πρωί έχουμε ψηφοφορία. Όσοι λοιπόν από εσά δεν Έχετε μαζί σας την ηλεκτρονική σας ε, κάρτα. Στείλτε κάποιον να σας τη φέρει. Ανακοινώσει του Πρόεδρου μου ζητήθηκε να επιτρέψω σε ένα συνεργείο να μπει γιατί θα γίνει ένα ντοκιμαντέρ για την προστασία των ε, δεδομένων έχουν λάβει μέρος και σε πολλές άλλες συνεδριάσεις Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Δεν υπάρχει λοιπόν αντίρρηση να μετασκοπήσουν τη συζήτησή μας για το συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή για την προστασία των δεδομένων. Να πω επίσης ότι έχουν αναβληθεί δύο σημεία από την ημερήσια διάταξη, συγκεκριμένα. Το σημείο 17, η ψηφοφορία της εκθέσεως μέρα δεν θα γίνει σήμερα η ψηφοφορία. Μιλάμε για τι θεωρήσει διαβατηρίων κατά τη δέληση εξωτερικών συνόρων. Αναβλήθηκε το σημείο αυτό. Αναβλήθηκε και το σημείο 19 τη έκθεση τη Ταβάρη, δηλαδή για την Ουγγαρία. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, συμφωνούμε προ την ίδια διάταξη. Επίση, θα πρέπει να εγκρίνουμε και τα πρακτικά τη τελευταία συνεδρίαση ε, μάλλον των τελευταίων συνεδριάσεων, 10 Δεκεμβρίου του 12, 26-27 Νοεμβρίου του 12, 20-21 Ιουνίου, 30-31 Μαου και 25-26 Απριλίου. Τα πρακτικά λοιπόν αυτά τα έχετε στη διάθεσή σα. δεν έχουμε πρόβλημα, νομίζω και μπορούμε να τα εγκρίνουμε. Περνάμε τώρα στο σημείο 4 την τρέχουσα κατάσταση δηλαδή των ανεξελίξη διοργανικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών. Έχουμε μαζί μας ε, τη Eurodac. Η ΛΥΜΠΕ ψήφισε για το θέμα Eurodac στις 17 Δεκεμβρίου. Στις 18 Δεκεμβρίου έλαβε χώρα ο πρώτος τρομερής διάλογος. Η κυρία Μακοβέ που είναι η θα μας αναφέρει τα σχετικά. Ποια δηλαδή ήταν η έκβαση του τριμερούς διαλόγου και τι περαιτέρω βήματα πρέπει να γίνουν. Κύριε Μακοβέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα σας πω ότι προέκυψε από την πρώτη συνάντηση του τριμερούς διαλόγου. Πρώτα απ' όλα ε, το blocking και marking των δεδομένων. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία ε, παροχής τελικών αποτυπωμάτων. Επίσης, τροπολογία στο άθρο 20 για την ανάγκη της ε, προεξάρουσας ε, προστασίας ε, της ασφάλειας και για την προστασία αυτών που έχουν ετηθεί διεθνούς προστασίας. Επίσης, τροπολογία την απαγόρευση μεταγωγών σε τρίτες χώρες ή διεθνών οργανώσεων και στοιχεία που έχουν να κάνουν περισσότερο με τις διμερείς επαφές με κράτη-μέλη. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Η Ιρλανδική Προεδρία εξέφρασε την πρόθεσή τη να προχωρήσει και αυτή γρήγορα για να υπάρξει συμφωνία επί Ιρλανδική Προεδρία. Μια τεχνική συνεδρίαση έλαβε τη χώρα στις 8 Ιανουαρίου. Η δεύτερη θα λάβει χώρα σήμερα. Ο επόμενο τριμερή ε, διάλογο θα προγραμματιστεί επίση σύντομα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη έκθεση με το πακέτο για τη διακυβέρνηση του Σέγγεν και έχουμε δύο συγητέ, ε, την κυρία Βέμπερ και τον κύριο Κοέλιο, που θα μα ενημερώσουν ε, για τον τεμεριδιάλογο ψηλού επίπεδου με τον κύριο Λουκά και με τον Επίτροπο Μάλμστρομ. Παρακαλώ. Κύριο Σκοέλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με την Προεδρία της Μάλτας, συνεργάστηκε πολύ στενά με το Κοινοβούλιο και έτσι καταφέραμε να φτάσουμε σε μια συνεννόηση. Τώρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν η Ιρλανδική Προεδρία θέλει να συνεχίσει με το θέμα αυτό και να φτάσουμε σε ολοκλήρωση. Αυτό που συμβαίνει, όπως γνωρίζετε, είναι ότι αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε ότι πρόκειται για θέμα συναπόφασης, ε, μάλλον συμφωνεί ότι είναι θέμα συναπόφαση. Το Συμβούλιο δεν θέλει να δώσει τη συναπόφαση στο Κοινοβούλιο. Εμεί προτείναμε μια εναλλακτική ε, να φτιάξουμε μια ρήτρα γέφυρα που συνδέει τον κώδικο Σέγγεν με τον μηχανισμό αξιολόγηση του Σέγγεν. Το Συμβούλιο δεν δέχεται την λύση αυτή και δεν έχει προτείνει κάποια εναλλακτική λύση. Εάν λοιπόν εμεί συμφωνήσουμε με την εκδοχή που μα, αν συμφωνούσαμε με την εκδοχή που μα υπευλήθηκε, θα σήμαινε αυτό τα εξή. Πρώτον, ότι θα εγκαταλείπαμε τη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου στην έγκριση του μηχανισμού αξιολόγηση του Σέγγεν Δεύτερον, θα εγκαταλείπαμε την ύπαρξη ενό μηχανισμού αξιολόγηση του Σέγγεν που να είναι πραγματικά ευρωπαϊκό. Τρίτον, δεν θα προστατεύαμε την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών. Και τέταρτον, θα αυξάναμε τις ιδιαιτερότητες που ήδη έχει ήδη το κάθε κρατός μέλος για την επανεισαγωγή δηλαδή νέων ε, συνοριακών ελέγχων. Θα σήμαινε δηλαδή ότι όλα αυτά αντίθετα με αυτά που υποστηρίζει το Ευρωκοινοβούλιο από πρώτη στιγμή. Ε, νομίζω λοιπόν πως ε, θα πρέπει να περιμένουμε. Δεν βλέπω κανένα, καμία προσπάθεια να γίνεται για να προσεγγίσουν το τις θέσεις μας. Και, αλλά θα πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία και στην Ελλανδική Προεδρία να δούμε πώς ξεπεράσουμε τη δύσκολη αυτή τη στιγμή. Ε, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την έκθεση. Καταλαβαίνουμε την κατάσταση. Φανταζόμαστε ότι η απόφαση που ελήφθη από την διάσκεψη των Προέδρων να μπλοκάρουν ολόκληρο το πακέτο μετά από την απόφαση του Συμβουλίου για αλλαγή της νομικής βάσης ε, για την ε, διακυβέρνηση του Σέγγεν δεν μπορεί να επιτευχθεί η Γενική Συμφωνία και θα πρέπει να ξαναρχίσουν εργασίες προς την, ε, υπό την Ιρλανδική Προεδρία, στην οποία ευχόμαστε να έχει επιτυχία όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά για όλα τα θέματα. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες και τα ζητήματα που διακυβεύονται εδώ. Αφού ακούσαμε τον κύριο Καοέλιο για το πακέτο αυτό, θα περάσουμε στο σημείο 5. και να θυμίσω ότι αυτή η συζήτηση γίνεται από μια ομάδα. Ναι, κύριε Ντόνομα, να έχετε ζητήσει το λόγο. Σας είδα, απλά να ανακοινήσω ότι τώρα πάμε στο σημείο 5 που είναι η προστασία των ατόμων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών ε, δεδομένων ελευθερία κίνηση των δεδομένων και γενικός κανονισμός προστασίας των δεδομένων. Έχουμε εδώ ένα δεύτερο στοιχείο του πακέτου για την προστασία των στοιχείων των δεδομένων. Έχουμε έναν κανονισμό. Πρώτος, το πρώτο θέμα αφορά τον κύριο Όλμπρεχτ, το δεύτερο τον κύριο Δρούτσα, ως εισηγητές και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Κομισιόν έχει παρουσίασει την πρόταση αυτή πέρσι, τέτοια εποχή. Τον Ιανουάριο του 2012 οι δύο εισηγητέ έχουν δουλέψει πολύ σκληρά μετά από διάφορες ε, ακροάσεις, παρουσιάσεις, ε, έγγραφα που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο και η Διακοινοβουλευτική Μικτή Επιτροπή συνεδρίασε τον Οκτώβριο του 2012 και αναπτύξαμε εκδεδομένη ανάλυση με κάποιες άλλες επιτροπές που έδωσαν γνωμοδοτήσεις, Ήτρε, Γιούρι και Ίμκο. Και οι δύο εισηγητές επί τη βάση της στενής του συνεργασίας και των παράλληλων διαδικασιών ε, τόνισαν την ανάγκη μιας ε, υιοθέτησης υπό την προσέγγιση πακέτου, όπως λέγεται. Και τώρα περιμένουμε από τους ηγητές να παρουσιάσουν το σχέδιο έκθεσης. Καταρχήν πάμε στον κύριο Άλμπρεχτ, λοιπόν, όπου μπορούμε και εδώ να δούμε την παρουσία των εκπροσώπων του κυρίου Μπουταρέλη, ο κύριος Μπουταρέλη που είναι εκπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκή, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Προστασία Δεδομένων ε, είναι στην αίθουσα νομίζω. Αλλά καταρχήν θα ακούσουμε του ηγητέ. Ο κύριο Άλμπρεχτ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και καλημέρα σε όλου. Έχουμε εδώ τα σχέδια έκθεσης ε, για τον κανονισμό και για την οδηγία για την προστασία των δεδομένων που ήταν αρκετά εκτεταμένη εργασία γιατί έπρεπε να εξετάσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν ήδη αρκετά ογκώδης. Μας πήρε αυτό αρκετές ε, συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους για να αναλύσουμε περί πρόκειται. καθώς επίσης και σε ποιο βαθμό οι συστάσει και οι απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν γίνει δεκτές και καθώς και ποιε αλλαγέ θα πρέπει να γίνουν στον κανονισμό ιδιαίτερα για το θέμα της ενίσχυσης των αρχών και των ορισμών που αποτελούν μέρος της πρώτης έκθεσης και των ετοιμάτων αυτής για τη διευκρίνηση και την ενίσχυση των μεμονωμένων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συγκατάθεση. Γιατί αυτό θα πρέπει να είναι ο γενικό κανόνα για την επεξεργασία των δεδομένων. Χρειάζονται σαφεί κανόνε και λιγότερε εξαιρέσει. Περισσότερη διαφάνεια δε. Και αυτό είναι και που προσπαθήσαμε να κάνουμε με, με το σχέδιο έκθεσης, να διευκρινίσουμε ιδιαίτερα στο άρθρο 6. Κατέστη σαφέ κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μα ότι εμεί ζητάμε ω κανονι... ως ε, νομοθέτες να θεσπίσουμε τους κανόνε, να μειώσουμε τον τεράστιο βαθμό ε, ε, πράξεων κατεξιοδότησης και εφαρμοστικών πράξεων στην έκθεση. Το κάναμε αυτό, έχουμε μειώσει στο μισό το ποσοστό των κατεξοδότηση και εφαρμοστικών πράξεων που έχουν αφαιρεθεί και έχουν ε, οριστεί περισσότερες και έχουμε έτσι φτιάξει περισσότερες διατάξεις και αυτά διατυπώνονται παράλληλα με τα όσα προτείνουμε στα έγγραφα εργασίας παλιότερα. Τα έγγραφα εργασίας όπως υπέδειξα και στην ε, παρουσίαση που σας έκανα με την ευκαιρία της προετοιμασίας τους και όπως σας ανέφερα στις επεξηγηματικές μου σημειώσεις υπάρχουν εδώ κάποιες προτάσεις στην έκθεσή μου που θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως βάση για τις επερχόμενες συζητήσεις γιατί θέλουμε ε, να φτιάξουμε μια ευρεία συνένεση για βασικά θέματα. Οπότε αυτό οφείλεται και στις ε, αλλαγές του μηχανισμού συνοχής. Ε, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι δεν θα πρέπει τελικά να είναι η Κομισιόν που αποφασίζει για τα DPAs αλλά μέσα στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει οι DPAs να βρίσκουν μια συμφωνία και το δικαστήριο να είναι το τελευταίο η τελευταία δυνατότητα προσφυγής για να δοθεί μια διερμηνία. Μια ερμηνεία. Ε, θέλουμε δηλαδή να δώσουμε περισσότερη νομική βεβαιότητα τους ε, όσους ασχολούνται με τα θέματα αυτά, από τη μια πλευρά δηλαδή τα άτομα και τις εταιρείες και από την άλλη τους πολίτες και τους πελάτες. Θεωρήσαμε πως οι κυρώσεις είναι πολύ σημαντικό τμήμα της έκθεσης ε, της Κομισιόν. Ήταν και κάτι το οποίο ζητήσαμε στην έκθεση το 2011. Ακολουθήσαμε λοιπόν την πρόταση της Κομισιόν αλλά είπαμε ότι αυτό θα πρέπει να κατευθυνθούν σαφώς από την αναλογικότητα. Η πρότασή μου είναι επίσης να, να απλοποιήσουμε τους κανόνες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ε, το... ο όγκος ελέγχου από πλευρά των ελεγκτών δεδομένων να περιοριστεί στα ατομικά δικαιώματα, δηλαδή ενημέρωση και δικαιώματα διαφάνειας. Και έτσι να μπορέσουμε να δείξουμε αυτή την τεκμηρίωση στις αρχές προστασίας δεδομένων όταν αυτό χρειάζεται. Επιπλέον, αναθέσαμε ευθύνες στους ε, ε, υπεύθυνου στους αρμόδιους προστασίας των δεδομένων που ορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όταν ορίζεται ένας τέτοιος ελεγκτής θα πρέπει να αναλαμβάνει και τις αντίστοιχες ευθύνες. Γι' αυτό πιστεύω πως αυτή η έκθεση καλύπτει πολλές ανησυχίες και απαιτήσει που εκφράστηκαν από διάφορες πλευρές και αυτό προσπάθησα και να κάνω κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου ώστε το Κοινοβούλιο να ακολουθήσει τις γραμμές των πρώτων συστάσεων είμαστε πρόθυμοι να εναρμονίσουμε την νομοθεσία να φτιάξουμε ένα σύνολο κανόνων που είναι ήδη ένα τεράστιο βήμα διότι πολλοί κόσμος στη ΣΥΠΑ είναι πρόθυμοι να το δεχτούν από τη στιγμή που υπάρχει ένα κοινό ε, πρότυπο, κοινέ προδιαγραφές σε υψηλό, υψηλό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, ω Κοινοβούλιο, εμεί θέλουμε να ακούσουμε όλου του ενδιαφερόμενου φορεί και αυτό κάναμε κιόλα. Εγώ ίδιο μπορώ να πω πώ έκανα τουλάχιστον 100 ε, επαφές με, διαφο με διαφορετικούς φορείς, κάναμε και ακροάσεις εδώ και μάλιστα μία συνάντηση κοινοβουλευτική ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και με ενδιαφερόμενους φορείς. Πιστεύω λοιπόν πως έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι διακυβεύεται εδώ. Εδώ έχουμε την πρώτη σύνοψη όπου περιλαμβάνονται και διάφορες συμβιβαστικές για τα όσα συζητήσαμε στις συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών και τώρα είμαι πολύ ικανοποιημένο ε, γιατί θα μπορέσω να έχω την δική σας ανταπόκριση και συμβολή, να δω τις τροπολογίες των διαφορών ομάδων. Συνεργαστήκαμε με τους συναδέλφους πάρα πολύ καλά. και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε ε, πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα σε όλες τις ομάδες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έχουν συνεργαστεί μαζί μου και έχουμε συγκεντρώσει τις διάφορες ιδέες καθώς και έχουμε συζητήσει σε μακρές συναντήσεις τις διάφορες ιδέες αλλά όλος ιδιαίτερος θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία που έκανε Πολύ εντατική δουλειά. Ήταν περίπλοκο να συνδυάσουμε τις διάφορες τροπολογίες. Είναι, ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και γι' αυτό και ευχαριστώ την γραμματεία. Υπάρχουν ωστόσο κάποια τεχνικά σφάλματα τα οποία διορθώσαμε τώρα. με ένα έγγραφο που αποκαλείται Εράτομ Σα ζητώ να το διαβάσετε. Υπάρχουν τροπολογίε που συνδέονται μεταξύ τους ή ε, ε, αλληλοδιορθώνονται. υπάρχουν και στοιχεία όπου δεν ερθώσαμε τις προτάσεις της Κομισιόν, δεν τις αλλάξαμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στη συζήτηση. Σας, σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή και τώρα να ακούσουμε τον κύριο Τρουτσά για την οδηγία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας καλή χρονιά Μια και ακολουθούμε αυτή την προσέγγιση του πακέτου, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε ο Γιάμ ο Γιάννα Αλμπρέχτη για το χρονοδιάγραμμα και για τις πρακτικές ε, διαστάσεις. Να επαναλάβω όμως τις ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν με εξαιρετικό τρόπο. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τη γραμματεία ασφαλώς. Και σε πιο προσωπικό επίπεδο επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μας στην πολιτική μου ομάδα και τους βοηθούς μας. Να τονίσω και πάλι αυτά που έχω επαναλάβει πολλές φορές ήδη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πετύχει ένα πολύ ψηλό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων και στόχος μας πρέπει να είναι να διατηρηθεί αυτό το υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πνεύμα λοιπόν αυτό, όλες οι τροπολογίες που προτείνονται στην έκθεση εξυπηρετούν το στόχο του να ενισχυθεί αυτό το επίπεδο προστασίας ε, σε συνάρτηση και με τον σχετικό κανονισμό και λαμβάνοντα υπόψη και τις λύσεις που προτείνονται. Να πω επίσης ότι η έκθεση ως σκοπό έχει να ενδυναμώσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τονίζοντας τα δικαιώματα του ατόμου, του ιδιώτη, δίνοντας ε, πιο μεγάλες δυνατότητες συντονισμού στις εθνικές αρχές προκειμένου να υπάρχει συντονισμός και διασυνοριακά. Να πω επίσης και να τονίσω, επειδή γίνονται κάποιες συζητήσεις σχετικά, αυτό θα το αναφέρω και λίγο παρακάτω, να σας ε, μιλήσω λοιπόν για το κατά πόσο είναι απαραίτητη ή όχι μια τέτοια οδηγία. Το επιχείρημα είναι ότι υπάρχει μια σχετική απόφαση του Συμβουλίου. Να σας πω όμως ότι αυτή η απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου δεν καλύπτει ένα συνεκτικό πλαίσιο από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, γιατί αναφέρεται μόνο σε διασυνοριακές περιπτώσεις. Δεν αναφέρεται σε εκπαραλλήλου υφιστάμενες διατάξεις μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών σε ό,τι αφορά τέτοια ζητήματα. Αυτό αποτελεί τη γραμμή που μας οδηγεί εμάς. Να ευχαριστήσω επίσης εκ νέου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο της. Καλωσορίζουμε τις προσπάθειες που έκανε για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προκειμένου να εναρμονιστούν και τα διαφορετικά ευρωπαϊκά συστήματα και θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματικά εξαιρετική η συνεργασία και επίσης να εκφράσω την ελπίδα το Συμβούλιο να ανταποκριθεί και αυτό στα καθήκοντά του σε ό,τι αφορά αυτή την προσέγγιση εν είδη πακέτου, την συνεκτική αυτή προσέγγιση και θα πω και δύο λόγια στο τέλος της παρουσίασης. Τώρα, εν συντομία, αν θέλετε επιγραμματικά, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις προτινόμενες αλλαγές στην έκθεση. Πρώτη αλλαγή. Κάθε εξαίρεση από την αρχή θα πρέπει να είναι σωστά δικαιολογημένη. Γιατί πρόκειται για ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου είναι θεμελιώδες δικαίωμα του. Και χρειάζεται πιο σαφή ορισμός των αρχών της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα στοιχεία διατήρησης ε, και φύλαξης δεδομένων, ενημέρωσης των στοιχείων, διατάξεις ελέγχου των δεδομένων σε περιπτώσεις που πρέπει να αποδεχτεί η συμμόρφωση με τους κανόνες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η ίδια γλώσσα, θεωρούμε, κατά το δυνατόν ασφαλώς, που χρησιμοποιείται και στον κανονισμό σε ό,τι αφορά τους ορισμούς. Επόμενο θέμα η επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει να είναι νόμιμη, δίκαιη και διαφανής σε ό,τι αφορά και τα άτομα που αφορά. Επίσης, τα δεδομένα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς που δεν συνάδουν με το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Επίσης, θα πρέπει να δικαιολογούν κάποιο στόχο. Και ο στόχος θα πρέπει να μην είναι δυνατόν να επιτευχθεί με άλλα μέσα. Επίσης, ένα σαφής ορισμός για το profiling. Αυτό έλειπε από την πρόταση για το profiling. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε την ίδια ευαισθησία και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα του profiling για τους πολίτες μας. Ύστερα, το Καθεστώ για την μεταφορά των δεδομένων σε τρίτε χώρε ήταν αρκετά δύναμο και δεν περιείχε όλες τις ασφαλιστικέ δικλείδε για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών των οποίων τα δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν. Άρα συμπεριλάβαμε και ένα καινούριο κεφάλαιο σχετικά. Και τέλος, να αναφερθώ στο ρόλο και στις εξουσίες των αρχών προστασίας των δεδομένων προκειμένου να ελέγχουν και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανόνες. Αυτά τα καθήκοντα θεωρούμε ότι δεν είχαν οριστεί με τον κατάλληλο τρόπο. Άρα θεωρούμε ότι δεν ήταν αρκετά σαφής η σαφή τα καθήκοντά τους. Αυτό το διορθώσαμε. Τώρα, Πρόεδρε, δύο λόγια να πω για να έχουν χρόνο και οι συνάδελφοι να κάνουν τα σχόλιά τους για τις εκθέσεις αυτές. Να πω δύο λόγια λοιπόν για την ε, προσέγγιση αυτή την συνεκτική, τη συνολική, το package approach. Να τονίσω ότι θεωρούμε ότι το, ο κανονισμός και η οδηγία αποτελούν πραγματικά ένα ενιαίο πακέτο, ένα ενιαίο σύνολο. Και αυτό ε, εξακολουθεί να ισχύει εντό του χρονοδιαγράμματο που έχουμε και για την υιοθέτηση και των δύο μέσων. Να σας υπενθυμίσω και πάλι ότι λάβαμε κάποια μάλλον απεσιόδοξα μηνύματα από τα κρατη στο Συμβούλιο που φαίνεται ότι διστάζουν αρκετά σε ό,τι αφορά την περαιτέρω εργασία για την ε, οδηγία. Στην Επιτροπή πρέπει να πω ότι έχουμε ένα καλό σύμμαχο και η Επιτροπός Ρέντινγκ δημόσια μας έχει υποστηρίξει και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει δηλώσει ότι ο κανονισμός και η οδηγία θα αποτελέσουν το ε, στοιχεία ενός ενιαίου πακέτου και να σας πω ότι σε επαφές με την Ιρλανδική Προεδρία τα μηνύματα ήταν αρκετά αισιόδοξα. Η Ιρλανδική Προεδρία μας ε, έδωσε το μήνυμα ότι θέλει να συνεχίσει η εργασία για την οδηγία και τώρα θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των κρατών μελών. Θα ήθελα να κλείσω τονίζοντας εκ νέου αυτή την συνολική προσέγγιση. Αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο τα νομοθετήματα αυτά και είμαστε διτεθειμένοι να λάβουμε ό,τι μέτρο χρειαστεί προκειμένου να πραγματοποιηθεί η υλοποίηση του πακέτου αυτού. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο, ευχαριστούμε τον κύριο Τρούτσα, σας ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης και φυσικά για το γεγονός ότι τονίζεται ότι θα πρέπει να τηρηθεί αυτή η αρχή που την θέσαμε εξ αρχής άλλωστε αυτή η συνολική προσέγγιση και η πρόταση κανονισμού και η πρόταση οδηγίας σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της αρχής αυτής. 15 μέλη έχουν ζητήσει το λόγο. Να σας πω ότι στις 11 έχουμε ψηφοφορία και ξέρετε πως πάνε οι ψηφοφορίες. Θα έρθουν κάποιοι συνάδελφοι που δεν θα έχουν έρθει μέχρι εκείνη την ώρα. Άρα αυτό θα πρέπει να το σεβαστούμε, θα ακούσουμε και τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Αν θέλετε, σας παρακαλώ να περιοριστείτε σε δύο λεπτά στις εισηγήσεις σας. Ασφαλώς το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε πολύ σημαντικά κεφάλαια ανοιχτά και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για το άσυλο, για το Σέγγεν. Για να ολοκληρώσουμε όμως τη συζήτηση μέσα σε μία ώρα, μιας και έχετε ζητήσει τόσο πολύ το λόγο, σας παρακαλώ, δύο-τρία λεπτά, δύο-τρία λεπτά ο καθένας, για να μπορέσουμε να ακούσουμε και την απάντηση των εισηγητών. Να δώσουμε καταρχά το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθότι αυτοί είναι και οι συντάκτες της πρόταση. Ίσως θα θέλετε να πείτε δύο λόγια πρωτού ξεκινήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω του εισηγητέ καταρχάς για τις πολύ χρήσιμες εκθέσεις τους. Γνωρίζουμε ότι οι εκθέσεις αυτές στηρίζουν την προσέγγιση της Κομισιόν για ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων στην Ευρώπη. Η Κομισιόν θεωρεί ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα ε, οδηγήσει σε μεγάλη συνένεση γιατί το υψηλό επίπεδο προστασία δεν είναι μόνο καλό για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη, για του πολίτε, αλλά είναι και καλό για να υπάρξει απαραίτητη εμπιστοσύνη για να μπορούν και οι επιχειρήσεις να καινοτομούν. και να υπάρχει εμπιστοσύνη από την πλευρά των πολιτών ότι γίνεται και ορθή χρήση των δεδομένων από τι επιχειρήσει. Δεν θεωρούμε τώρα ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ του υψηλού επίπεδου προστασία αφενό ε, και τη ε, τήρηση των κανόνων για την εθνική επεξεργασία φετέρου. Υπάρχει αποτελεσματική επιβολή τη νομοθεσία. Θέλω να ευχαριστήσω του συζητητέ και να του ευχαριστήσω και για κάτι ακόμη, γιατί κατέβαλαν προσπάθεια να συνεργαστούν με του κοιόδε συζητητέ ε, και με όλε τι πολιτικέ ομάδε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προφανώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να προχωρήσουμε ομαλά μέχρι την ολοκλήρωση αυτού του φακέλου. Προσβλέπουμε λοιπόν και εμείς στη διατήρηση αυτής της καλής συνεργασίας με τους εισηγητές και με όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν επίσης φυσικά και θα βοηθήσει για την εξομάλυνση της συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Αυτό το οποίο επιθυμούμε το είπε και ο εισηγητή Αλμπριχτ, είναι να επιτευχθεί ταχεία πρόοδο και περιμένουμε να δούμε την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο τον Απρίλιο. Πιστεύουμε ότι η Ιρλανδική Προεδρία πραγματικά ε, καταλαμβάνει επιτυχημένες προσπάθειες για να προχωρήσουμε τάχιστα και σε επίπεδο Συμβουλίου με αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και φυσικά και θα συνεργαστούμε επικοδομητικά και στη συνέχεια μαζί σας για την ολοκλήρωση θέματος. Ο επόπτη ε, προστασία δομών, κ. Μπουταρέλη, είχε να πει κάτι. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε και εμείς ως όργανο σε αυτή την πρώτη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναγνωρίσω ότι μετά από ένα έτος τατικών ε, συναντήσεων, σεμιναρίων, εργαστήρων κτλ. Δεν ήταν τόσο απλό για τους δύο να βρουν τη σωστή ισορροπία και να ικανοποιήσει ταυτόχρονα και όλες τις προσδοκίες. Μας εντυπωσιάζει λοιπόν η τεράστια προσπάθεια που αποσκοπεί στην εξισορρόπηση των διαφορετικών μεταξύ τους και κάποιες φορές αντικρουόμενων συμφερόντων των εμπλεκομένων. Εμείς από την πλευρά του υπότιτλου προστασίας δεδομένων σημειώνουμε ότι τον Οκτώβριο τα περισσότερα από όσα ε, είχαμε εκφράσει τη γνωμοδότησή μας του Μαρτίου ε, στα τρία ε, έγγραφα εργασία που δημοσιεύτηκαν, παραλαμβάνω τον Οκτώβριο, λαμβάνονται υπόψη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι δύο πολύ μελλοντικέ εκθέσει ε, ακολουθούν την ίδια προσέγγιση. Έχουμε ξεκινήσει μια ανάλυση σε βάθο, η οποία θα απαιτήσει βέβαια και μια προσεκτική αξιολόγηση των εγγράφων αυτών. Θα ήθελα όμω να πω δύο λόγια, τονίζοντα καταρχά ότι οι δύο εκθέσει φαίνεται όπω ε, είπε και ο Πολ Νέμι, φαίνεται να βασίζονται και στην Κομισιόν, στην Κομισιόν και στο σχετικό τη έγγραφο. Βέβαια σε κάποια σημεία διαφοροποιούνται. Εμείς στηρίζουμε τη διαδικασία να θεωρηθούν πακέτο αυτά τα δύο νομικά μέσα. Η προσπάθεια των δύο συγγητών για καλύτερη ευθυγράμμιση αυτών των δύο μέσων, για ενίσχυση της οδηγίας, ε, μας βρίσκει σύμφωνο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κανονισμό, Καταρχήν, συμφωνούμε και στις 10 βασικές γραμμές τις οποίες ε, ανέφερε ο εισηγητής Άλμπρεχτ ε, στη συνδεξιτή που έδωσε. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κανονισμό, ακριβώς τον ίδιο κανονισμό, εκτιμούμε την πρόθεση να διευκρινιστούν ορισμένες διατάξεις για τα δικαιώματα των ατόμων, για την διαφάνεια της επεξεργασίας, για την αρχή της αρχής lead authority της αρχής που έχει τον πρώτο λόγο αλλά δεν θα θεωρήσουμε ότι έχει την αποκλειστικότητα αλλά θα πρέπει να συνεργάζεται και με άλλες υποπτικές αρχές. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν βελτιώσεις και σε ό,τι αφορά ε, τον σχετικό μηχανισμό, τις διαδικασίες, επιλεκτικές διαδικασίες που τον ενεργοποιούν ή την απαραίτητη ευελιξία, τα πιο ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα που είναι απαραίτητα για την έγκριση και των γνωμοδοτήσεων του επόπτη προσέσεις δεδομένων. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξουσίες της Κομισιόν, την ε, επιλεκτική διαδικασία, εξουσιοδότηση, εφαρμοστικές, τελεστικές πράξεις, ευελιξία, διοικητικών κυρώσεων κτλ είναι πολύ καλές σχετικές ε, προσεγγίσεις, αλλά και σε ό,τι αφορά την ε, μείωση του διοικητικού βάρους. Θέλουμε να έχουμε επιτυχημένη και αποτελεσματική προστασία των θεμελιών δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν ε, καλή η βάση εργασίας αυτή των δύο αυτών εγγράφων. Τώρα, Βλέπουμε επίση ότι υπάρχει προσπάθεια αύξηση του επίπεδου προστασία των δεδομένων ε, με την εισαγωγή κάποιων θετικών στοιχείων στο πλαίσιο τη λεγόμενη αρχή τη ευθύνη ή λογοδοσία, κάτι το οποίο έλειπε από την αρχική πρόταση οδηγία για τη ρύθμιση ανταλλαγή ε, πληροφοριών μεταξύ αρχών επιβολή νομοθεσία, ιδιωτικού τομέα ή βελτιώση των διατάξεων για τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες. Εν κατακλείδη λοιπόν, εκτιμούμε την δέσμευση και αφοσίωση που δείχνουν δύο συγκητές για την ευθυγράμμιση των δύο προτάσεων. Είμαστε διαθέσιμοι σε όλους σας βέβαια και για περαιτέρω συνεργασία και θα συνεχίσουμε από πλευράς μας να αναλύουμε ε, τα στοιχεία και όπου χρειαστεί θα κάνουμε και επίσημες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Πουταρέλ και τώρα ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα δώσω πρώτα το λόγο στους ε, σκιώδεις εισηγητές. Δεν ξέρω αν θέλει να ξεκινήσει ο κύριος Σάλβαρο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα γερμανικά. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα να μιλάμε τη μητρική μας γλώσσα και να πω ότι, ότι πέρα από κάθε αμφιβολία σε ό,τι αφορά την πρόταση του κανονισμού υπάρχουν σημεία κριτικής αλλά είναι αξιόλογο το ότι ο συνάδελφος Άλμπρεχτ κατάφερε με τόσες πολλές σελίδες να επηρεάσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και με δημιουργικές ιδέες να συμμετάσχει στην συζήτηση αυτή και θεωρώ ότι ήδη έχει αφήσει τη σφραγίδα του το αποτύπωμά του στη συζήτηση αυτή. Κάποια στοιχεία ωστόσο θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητηθούν. Κοιτώντα ε, φυσικά ότι δεν μπορούμε να πει σε λεπτομέρειες εμεί και δεν έχουμε πολύ χρόνο, θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή θα πρέπει να προσανατολίζεται στο ποιοι είναι οι σκοποί και ποια είναι τα καθήκοντα της προστασίας των δεδομένων. Ο έλεγχος. Ο έλεγχος είναι, είναι κάτι που μπορούμε να το πετύχουμε μόνο όταν υπάρχει ασφάλεια απόφασης. Είναι δύσκολο λοιπόν να περιοριστεί υπερβολικά αυτή η δυνατότητα λήψης αποφάσεων του ατόμου. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τον, την αλλαγή του ορισμού του ατόμου και των ε, δε, προσωπικών δεδομένων. Ουσιαστικά τα πάντα α, μπορούν να καταστούν προσωπικά δεδομένα. Για την τροπολογία δηλαδή 4 για το άρθρο 4.1 αλλά δεν θα πρέπει να παραφορτώσουμε την προστασία των δεδομένων προκειμένου να ε, μην είναι εφαρμοστέα στην τελική ανάλυση. Θεωρώ ότι κάποιες αλλαγές που είχαν καλό σκοπό, όπως το άρθρο 6, το άρθρο 15, θεωρώ ότι αποτελούν παρεκκλήσεις και παραθυράκια, αν θέλετε, για μη αποσκοπούμενες ε, και εκμετάλλευσης των προσωπικών δεδομένων. Για την 59 και 64 θεωρώ ότι αφορούν πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσα κακά, αλλά θεωρώ ότι πράγματα που έχουν ρυθμιστεί στην οδηγία δεν χρειάζονται να τα ρυθμίζουμε και στον κανονισμό και σε ό,τι αφορά τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι που πολλοί συνάδελφοι αναγνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει αυτά που οφείλει να κάνει. Υπάρχουν αρμοδιότητες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το θέμα μάλλον δεν είναι να μεταφέρουμε αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το ε, Συμβούλιο ε, Εποπτείας των Προσωπικών Δεδομένων, γιατί ουσιαστικά μεταφέρουμε από μία μη από ένα μη νομιμοποιημένο όργανο σε ένα άλλο τις ε, αρμοδιότητες αυτό, αυτές. Και αυτό δεν δημιουργεί νομική βεβαιότητα αν ένας νόμος υπόκειται διαρκής τραποποίησης, δεν βοηθάμε κανέναν, ούτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτε τις μεγάλες επιχειρήσεις, ούτε κανόναν. Άρα η νομοθεσία θα πρέπει να ρυθμίζει ό,τι είναι να ρυθμίσει και αν υπάρχουν ανάγκες να υπάρξει τροποποίηση, να γίνει αυτό μέσω του Κοινοβουλίου. Το ίδιο ισχύει όταν ρυθμίζεται κάτι σε μια άλλη οδηγία και μάλιστα με τρόπο που φαίνεται ότι λειτουργεί, γιατί θα πρέπει να τα ρυθμίσουμε αυτά εκ νέου σε ένα κανονισμό. Αυτό δεν το καταλαβαίνω και θα πρέπει να το σκεφτούμε σε ό,τι αφορά τον ε, υπεύθυνο για την ε, προστασία των δικαιωμάτων θα πρέπει να έχει να φτάνει με την εξουσία, με το power όπως αναφέρεται στα αγγλικά, της ε, προστασίας των δεδομένων. Και επίσης καθοριστικό είναι, ξέρω ότι θέλετε να τελειώνω, αλλά είναι κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε αυτά. Τα τεχνικά πρότυπα. Θεωρώ ότι και αυτά δεν μπορεί να τα ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το ορίζουν και θα πρέπει να το ορίζουν αυτοί που συμμετέχουν και καθορίζουν την αγορά. Ο κανονισμός, θεωρώ λοιπόν, πρέπει να ορίσει το τι θα πρέπει να ισχύει ως νόμος και όχι το πώς θα πρέπει να επιτευχθεί αυτό. Αυτό είναι καθοριστικό. Οι μεμονωμένες προδιαγραφές ή λεπτομέρειες θεωρώ ότι δεν μας βοηθούν και συγγνώμη που μακρηγόρησα αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν. Thank you, Mr. Alvaro. Σας ευχαριστώ κύριε Αλβαρό. Είπα δύο-τρία λεπτά από καθένας. Παρακαλώ, όχι πέντε. Αλλιώς θα βρεθούμε στη συνήθεια ενοχλητική κατάσταση όταν πρέπει να ψηφίσουμε σε 11 να μην έχουν μιλήσει όλοι. Ο επόμενος ομιλητής Κιώδης για το ΕΛΚ παρακαλώ. Κύριε Φως, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να παραπονεθώ λίγο για το, τη διαδικασία που ακολουθούμε. Πώς μπορούμε να ασχοληθούμε μέσα σε δύο λεπτά με δύο νομοθετικές πράξεις. Σε ένα τέτοιο θέμα, σας παρακαλώ, μη μας περιορίζετε. Να σας πω, κύριε Φως, το εξής. Φυσικά και καταλαβαίνω, λέει ο Πρόεδρος, και ξέρω ότι πάντα προσπαθούμε να επιτύξουμε μια ευελιξία. Δεν ναι, θα κλείσει εδώ η συζήτηση. Εδώ ξεκίνησε η παρουσίαση της έκθεσης. Αν ε, θεωρηθεί απαραίτητο, θα υπάρξει και συνέχεια της συζήτησης αυτής στην επόμενη τακτική συνάντηση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. 21 και 22 Ιανουαρίου. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο συζητήσεων όπως σας είπα όμως, η κατάσταση ξέρετε ποια είναι. Όταν ξεκινάει η ψηφοφορία, μπαίνουν κάποιοι συνάδελφοι που έρχονται μόνο για την ψηφοφορία και διαμαρτύρονται, άμα δεν είμαστε έτοιμοι. Να δείξουμε με ευελιξία, αλλά σας παρακαλώ μιλήστε και μην διαμαρτύρεστε. Ευχαριστώ πολύ και με ικανοποίησατε που το είπατε αυτό ότι θα υπάρξει και συνέχεια της συζήτησης. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την ανοιχτή συνεργασία αγαπητοί εισηγητές και ασφαλώς δεν μπορούμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να τα συζητήσουμε και να τα αξιολογήσουμε όλα. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο κόσμος στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε. Και σωστά είπε ο συνάδελφος Άλβαρο ότι ο πολίτης στην ε, εποχή του ίντερνετ θέλει καταρχάς προστασία των προσωπικών δεδομένων του και της ιδιωτικής του σφαίρας, αλλά παράλληλα υπηρεσίες, προσφορές που δεν έχουν το σχετικό κόστος και για τις οποίες πρέπει να διαθέσει τα δεδομένα του. Άρα δεν μπορεί να είναι εξαιρετική αυτή η προστασία των προσωπικών δεδομένων, υπερβολικά αυστηρή, γιατί αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει και ε, μειονεκτήματα για τον πολίτη. Πιο ακριβά δάνεια, λιγότερες προσφορές και το καθεξής. Άρα χρειαζόμαστε μια ισορροπία προς τη σωστή κατεύθυνση οδεύει η έκθεση, αλλά πότε το έχει πετύχει αυτό, θεωρώ, ακόμη. Και τώρα σας τα αναφέρω όλα αυτά επιγραμματικά. Δυστυχώς, μετά από μια πρώτη αξιολόγηση, μου αρέσουν πολύ τα εξή. Σε ό,τι αφορά τον υπεύθυνο προστασία των επιχειρηματικών δεδομένων. Αναλαμβάνουν και αυτοί οι ευθύνε. Αυτό είναι θετικό στο πνεύμα της αυτορύθμισης μπορούμε να πάμε και λίγο παρακάτω. Το right to be forgotten περιορίζεται με ρεαλιστικό τρόπο. Ίσως θα μπορούσαμε σε δύο φορά το δικαίωμα διαγραφής και το δικαίωμα αυτό το right to be forgotten να συζητήσουμε περαιτέρω για τη μεταφορά των δεδομένων θεωρώ ότι τα αναφέρεται σωστά. Ίσως θα έπρεπε να συμπεριληφθεί και το επιχειρηματικό απόρριτο καλό το ότι συμπεριλαμβάνονται και τα ανώνυμα δεδομένα. Συμφωνώ και με τον περιορισμό των τελεκριτάκτης των ε, πράξεων κατά Αυτά που δεν με ικανοποιούν απαραίτητα θεωρώ ότι ο ορισμός των προσωπικών δεδομένων, όπως είπε και ο κ. Άλβαρο, καλό θα είναι να εισαχθούν αυτά τα ε, αν θέλετε, ανωνυμοποιημένα στοιχεία. Η τροπολογία 105 μου φαίνεται αρκετά αντιφατική. Η προτανόμενη, ε, προτινόμενη λύση για το άρθρο 7 παράγραφος 4 θεωρώ ότι είναι προβληματική. Το νόμιμο συμφέρον είναι καλό, καλή είναι και η προσέγγιση με τα παραδείγματα, αλλά και εκεί θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και μήπως περιορίζει τις δυνατότητες της οδηγίας. Δεν υπάρχουν ρήτρες για τους ομίλους σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση για τα στοιχεία που αφορούν την υγεία των ιδιωτών. Αυτά μόνο για τον κρονισμό και για την οδηγία έχω πάρα πολλά στοιχεία, αλλά ίσως καλύτερα να τα συζητήσω με τον ε, εισηγητή κατηδίαν ή στην επόμενη ευκαιρία που θα έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κύρκοπ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ θα είμαι πολύ γενικόλογος και σύντομος, γιατί με ανακούφισε ότι άκουσα πως θα κάνουμε πιο εις βάθος ε, συζήτηση που πιστεύω ότι είναι απαραίτητη εδώ και όχι μόνο τη σημερινή συζήτηση που, βασικά είχαμε προειδοποιήσει πριν δύο μέρες για μια έκθεση που είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Επίσης θα ήθελα να δούμε στις 27 Φεβρουαρίου μήπως ε, την καθυστερήσουμε κάπως την εξέταση γιατί πάλι θα είναι δύσκολο για μας να δούμε όλες τις απαραίτητες τροπολογίες και την προπαρασκευαστική εργασία που πρέπει να κάνουμε μέχρι τις 27. Επίσης να πω ότι συμφωνώ με την ε, υπαρξή νομοθεσία περί ε, προστασίας των δεδομένων, Όμω ξέρουμε πω αυτή δεν εφαρμόζεται ε, με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση. Και θα πρέπει επίση να ενημερωθεί, γιατί ο κόσμο κινείται πολύ γρήγορα. Και ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε μέχρι στιγμή. Αυτό που χρειάζεται φυσικά είναι σαφείς και συνεπεί κανόνες και υποχρεώσεις που να εφαρμόζονται σωστά. Αλλά επίση θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε σε αυτή μα την προσπάθεια να εξορροπήσουμε τα συμφέροντα όχι μόνο των καταναλωτών αλλά και τη ε, βιομηχανία μας γιατί το διοικητικό κόστος ε, ε, είναι σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως που αποτελούν τη βάση του, της μελλοντικής επιτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε την ανάγκη αυτής της μέρημνας να μην είναι εξαιρετικά λεπτομερής αυτή η έκθεση που θα μπορούσε εξάλλου και να ξεπεραστεί πολύ γρήγορα από τη στιγμή που συνεχίζονται οι πολύ γρήγορες αλλαγές. Επίσης θέλουμε να προσέξουμε για τον αριθμό των κατοξιδότησης ευθυνών της προς την Κομισιόν, οι οποίες κανονικά θα πρέπει να ανατεθούν στις ε, τοπικές, εθνικές αρχές μάλλον κάθε φορά, γιατί αυτές αντιμετωπίζουν επιτόπου τα προβλήματα. Επίση, ε, είμαστε κατά της περάτασης ε, των περιόδων, των περιόδων κοινοποίησης. Οι αρχικές ήταν, προθεσμίες ήταν πολύ στενές και μη καθόλου πρακτικές. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που έχω να πω αυτή τη στιγμή, Πρόεδρε. Ε, ε, δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες. Είναι πολύ σημαντικό βήμα για να προχωρήσουμε με την ψηφιακή ενιαία αγορά και να αυξηθεί το διεθνές εμπόριο, αλλά και οι σχέσεις μας με άλλα μέρη του κόσμου, ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ και τις μελλοντικέ μας σχέσεις τέτοιου τύπου. Προστασία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών δεν είναι δύο αντιφατικές έννοιες, θα έπρεπε να είναι απόλυτα συμβατές μάλιστα. Και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να μην πνίξουμε την καινοτομία και την ανάπτυξη και να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι και αν φτιάξουμε τελικά εδώ, να μένει στην ιστορία, και, αλλά και να είναι και βιώσιμο για τουλάχιστον ακόμα 15 χρόνια, ώστε να μην χρειάζεται διαρκώς να επιστρέφουμε στο θέμα αυτό και στις επιπλοκές που θα προκύπτουν από αυτό. Τέλος να πω πως είναι πολύ τεχνική η έκθεση. Πολλή δουλειά έχει γίνει μέχρι στιγμής για αυτήν. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε θετικά και είμαι βέβαιος πως τελικά θα φτάσουμε συμβαστικές αποδεκτές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ η κυρία Ιντουφέλτ που είναι η σκιώδης, η σκιώδης για έναν από τους ε, φακέλους. Ε, την οδηγία για την προστασία των δεδομένων. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους δύο εισηγητές που έκαναν τρομερή και όχι και πολύ εύκολη δουλειά ε, που μόλις ξεκίνησε μάλιστα οι δύο εκθέσεις αντικατοπτρίζουν τις συζητήσεις που κάναμε τον τελευταίο χρόνο, τον περασμένο χρόνο όλοι γνωρίζουμε πως ε, τα λόμπι για αυτό το φάκελο είναι πολύ έντονα ε, και αυτό που είναι επίσης ενδιαφέρον είναι ότι όλες αυτές οι ομάδες πίεσης έχουν αντιφατικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Είπαμε επίσης εξ ότι όσοι θα πρέπει να, να δεχτούν την καινοτομία ε, και είμαι, γνωρίζω πως το Κοινοβούλιο θέλει να υπάρχει ένα μόνο μέσο το οποίο θα ισχύει για τη ε, προσωπικά δεδομένα. Δυστυχώς αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό. Θα προσπαθήσουμε ωστόσο να ευθυγραμμίσουμε τα μέσα ώστε να φτάσουμε σε ένα ενιαίο επίπεδο προστασίας. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η οδηγία θα πρέπει να δεχτούμε ε, και την εξαιρέσεις ε, στον κανόνα και πραγματικά εγώ θα ήμουν αντίθετη οποιασδήποτε προσπάθειας ε, του Συμβουλίου για να περιληφθούν εδώ οποιασδήποτε κανόνες που δεν ασφορούν την επιβολή του νόμου και την ασφάλεια. Γιατί πιστεύω πως το Συμβούλιο προσπαθώντας να καθυστερήσει τις συνομιλίες ε, για αυτή την οδηγία ε, δρά τελείως ανεύθυνα. Ενεργεί τελείω ανεύθυνα, γιατί το σωστό επίπεδο προστασία δεν είναι εμπόδιο στη χρήση των δεδομένων, είναι προϋπόθεση για τη χρήση αυτών. Στην ε, συνεργασία της αστυνομίας και της δικαιοσύνης η απουσία ε, νόμων περί προστασίας δεδομένων είναι εμπόδιο και έχουμε δει πολλά παραδείγματα για το πώς οι εγκληματίες ξεφεύγουν επειδή ακριβώς δεν υπάρχει μια κατάλληλη βάση για την ανταλλαγή ε, στοιχείων σύντομα για κάποιες από τις συγκεκριμένες προτάσεις για τις εκθέσεις και για τις δύο εκθέσεις. Με χαρά είδα ότι οι παράγραφοι που αφορούν ε, τις μεταφορές τρίτων χωρών έχουν επανέλθει. Ε, νομίζω πως θα πρέπει να εξετάσουμε στενότερα όλες τις λεπτομέρειες γιατί φαίνεται ότι οι, αυτές οι, παραγρα... παράγραφοι είναι πολύ καλές και το γεγονός ότι το μέγεθος της εταιρείας δεν είναι το σημαντικότερο. Ε, σημαίνει απλοποίηση η οδηγία, θα πρέ... όπως σας είπα, θα πρέπει να παραμείνει εξαίρεση στον κανόνα. Με χαρά είδα ότι και οι δύο εισηγητές αναφέρονται σε άλλες ε, οργανισμούς της Ένωσης που καλύπτονται από χωριστούς κανόνες αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να στοχεύσουμε σε ένα νέο, εναρμονισμένο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Νομίζω πως χρειάζεται περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των κανόνων, ας πούμε, για την προστασία για στόχους ε, δημόσιου συμφέροντος. Ε, εντάξει, ωραίο ακούγεται, αλλά πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι περί τίνος πρόκειται. Και έπειτα να κάνουμε και μια εξέταση όσον αφορά τις εξαιρέσεις. Ο κανονισμός θα μπορούσε να είναι λίγο πιο γενναιόδωρος εκεί. Αυτά Έχω να πω για την ώρα, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κυρία Ιντεβέλτ. Ο κύριο Ταβάρε, σειρά σας. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ένα σημείο έχω για την κάθε έκθεση. Ξεκινώ με την έκθεση του Γιάνν Άλμπρεχτ, που είναι και ένας από τους καλύτερους μου φίλους εδώ στο Κοινοβούλιο και τον θαυμάζω ως βουλευτή. Διάβασα την έκθεσή του και νομίζω ότι υπάρχουν ε, πολύ καλά στοιχεία σε αυτήν. Βλέπουμε και με τις τροπολογίες ότι αυτό που κάνει η έκθεσή του είναι να εξορροπήσει την εξουσία μεταξύ θεσμών και απλού πολίτη. και θεσμών και μεγάλων επιχειρήσεων απέναντι στον πολίτη, γιατί θέλουμε να υπάρχει μια συμμετρία στην παροχή πληροφοριών. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο που αφορά ακριβώς αυτό το σημείο, την συμμετρία της ενημέρωσης των πληροφοριών. Έχουμε και τις πολιτικές περιπροστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα βλέπουμε σε διάφορες ιστοσελίδες ε, όταν ζητούνται προσωπικά δεδομένα. Και όλες αυτές οι διατάξεις που δεν τις διαβάζει κανένας είναι και μακροσκελής και πολύπλοκες και δεν μπορεί να τις καταλάβει ένας απλός πολίτης. Χρειάζεται δικηγόρος για να στα εξηγήσει όλα αυτά. Ο απλός πολίτης ε, βέβαια σίγουρα δεν έχει μια ομάδα δικηγόρων στη διάθεσή του. Ο Γιάννα Άλμπρεχτ λοιπόν με την τροπολογία 71 ζητά κατεξοδότηση πράξη από την Κομισιόν ε, για να έχουμε ένα ε, ενοποιημένο μοντέλο για την ε, παροχή πληροφοριών. Και αντί να χρειάζεται κανείς να διαβάσει μπαίνοντα στο ίντερνετ ένα συμβόλαιο που δεν το καταλαβαίνει, να έχει κάποια τυποποιημένα εικονίδια. Και μέσα σε δευτερόλεπτα να μπορεί με τον τρόπο αυτό να καταλάβει πού ε, πηγαίνουν τα δεδομένα του πολίτη και με ποιες προποθέσεις, από ποιου όρους, πόσες μέρες θα διατηρήσει στο ιστοσελίδα τα στοιχεία του, ε, πού μπορεί να τα διαθέσει κτλ. κτλ. Εγώ θα επεξεργαστώ και κάποιες τροπολογίες σχετικά με το σημείο αυτό για να βοηθήσω να οριστεί καλύτερα το πλαίσιο αυτό για την κατεξουσιοδότηση πράξη και η σχετική προθεσμία. Και αν προσπαθήσουμε χωρί κατεξουσιοδότηση πράξη να πετύχουμε αυτό που θέλει ο Γιάννη Άλμπερτ, θα ήταν ίσω καλύτερο. Βέβαια δεν είναι κάτι ε, που το ακούμε για πρώτη φορά και ο Αλεξάνδερ Άλβαρ και άλλοι το έχουν ε, αναφέρει. Θα μπορούσαμε ίσως κάποιοι συνάδελφοι λοιπόν να συνεργαστούμε για να επεξεργαστούμε μια σχετική πρόταση και βέβαια να συντονιστεί τον εισηγητή μας. Για τον συνάδελφο Δρούτσα Θέλω να πω ότι διάβασα τα σχόλιά σας στην ετολική σας έκθεση σε ό,τι αφορά το profiling και την ανάγκη να υπάρξει μια ισορροπία ώστε να μην είναι δυνατόν αυτό το profiling να μεταλλαγεί ε, και να μπορεί τελικά ε, να χρησιμοποιηθεί ώστε να παγιδεύει κατά κάποιο τρόπο κάποια άτομα ε, δίνοντας κάποια χαρακτηριστικά ε, ιονή υποπτή συμπεριφοράς. Μήπως θα ήταν καλύτερο να μην είναι νόμιμο αυτό το profiling. Ε, δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να διευκρινίσετε το θέμα αυτό και να σας ευχαριστώ και τους δύο γιατί έχετε εργαστεί πολλές ώρες για τις εκθέσεις σας. ο κύριος Δίκστρα είναι ο επόμενος ομιλητής. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. το γεγονό ότι αντιμετωπίζουμε πολλά θέματα που αφορούν την προσωπική των δεδομένων δεν το αρνείται κανείς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και στον κανονισμό αυτό ε, θέλουμε να ασφαλίσουμε ακριβώς τα προσωπικά δεδομένα. Τρεις παρατηρήσεις έχω να κάνω. Καταρχάς, κατά πόσον έχουμε κοιτάξει επαρκώ το θέμα της αρχής της επικουρικότητας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή που απαραίτητος θα πρέπει να συντονίσει την προσπάθεια. Τα κράτη-μέλη δεν είναι ανίκανα εξόρισμου για να ορίσουν τους σχετικούς κανόνες στον τομέα αυτό και η συνθήκη αναφέρει την εναρμόνιση της νομοθεσίας αν είναι αυτό απαραίτητο για την ενιαία αγορά και τη λειτουργία της. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν αποτελεί επαρκή ε, αιτιολογία. Δεύτερη παρατήρηση ένα ενιαίο σύνολο ε, κανονισμών και ρυθμίσεων θα λειτουργήσει. Θεωρώ ότι ο κανονισμός δεν ε, τα καταφέρνει γιατί δεν ρυθμίζει μόνο το τι θα πρέπει να ρυθμιστεί αλλά και το πώς θα πρέπει να ρυθμιστεί. Αυτό το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές και οι κανόνες προστασίας ισχύουν ε, για όλους τους οργανισμούς κάποιας, κάποιου μεγέθους αυτό σημαίνει ότι σε κάποιε περιπτώσεις θα υπάρχει μεγάλο άχθος γραφειοκρατικό για κάποιε επιχειρήσεις χωρίς να ωφελεί αυτό τον πολίτη και θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλη η ωφέλεια. Και τρίτο και πιο σημαντικό θα πρέπει να τονίσουμε πιο πολύ την ιδιοκτησία των δεδομένων. Επιτρέπεται στον ψηφιακό κόσμο να ακολουθούνται ακόμα και παιδιά ένα ψηφιακό κόσμο που αυξάνεται διαρκώς. Όλα τα email που γράφει κανείς, ε, ό,τι διαβάζει κανείς, κάθε φωτογραφία που στέλνει, όλα αυτά ε, μένουν και δεν διαγράφονται. Και αυτά αποτελούν και αντικείμενο εμπορίας. Και έχουν οικονομική αξία. Θα πρέπει να συζητήσουμε όμως και κατά πόσο ε, είναι λογικό να μπορεί κανείς να είναι ανώνυμος στο ίντερνετ. Το γεγονός ότι θα πρέπει τα παιδιά να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε για το δικαίωμα να μπορεί να ξεχαστούν κάποια στοιχεία. Τα λόμπι ε, δεν συμφωνούν, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει περαιτέρω συζήτηση και θεωρώ ότι η συζήτηση θα πρέπει να έχει και κοινωνικό χαρακτήρα γιατί θεωρώ ότι θα είναι μεγάλος ο αντίκτυπος για τη χρήση των αγορασμένων προσωπικών δεδομένων, όπου ο πολίτης ε, έρχεται αντιμέτωπος με μια εταιρεία με την οποία δεν έχει έρθει ο ίδιος σε επαφή. Έχει αυτό να κάνει με το δικαίωμα να ξεχαστεί κανείς. Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να μα οδηγήσει σε μια λογική και καλή χρήση των προσωπικών δεδομένων αυτών και αυτό θα πρέπει να εξαρτάται και από τον ίδιο το πολίτη, κατά πόσον θέλει να βεβαιωθούν τα στοιχεία αυτά. Κυρία Αναχέντα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον εισηγητή, γιατί ε, πολύ καλή έκθεση. Θα ήθελα στα δικά μου σχόλια να αναφερθώ στην έκθεση για το γραφείο για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αναφέρονται όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και θεωρώ ότι αυτό θα αποτελεί ένα καλό τρόπο να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων αυτών. Να θυμόμαστε άλλωστε ότι κάποια από τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι σχετικά και θα πρέπει να τα δούμε σε συνάρτηση με άλλα δικαιώματα άρα, στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι κάποια δικαιώματα, κάποια μάλλον ε, ε κάποιες έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των παιδιών που χρήζουν ιδιαίτερες προστασίες. Και υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις με τη συνθήκη για τα δικαιώματα του παιδιού που έχουν ε, υπογράψει όλα τα κρατημέλη και Πρέπει να πω ότι οι συγητές έχουν συμπεριλάβει και πολλά καλά στοιχεία σε ό,τι αφορά την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και των δικαιωμάτων του ατόμου. Έχω θέσει κάποια, κάποια ερωτήματα σχετικά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μου έχουν απαντηθεί επαρκώ ε, στο άρθρο 80 θεωρώ ότι τίθονται αρκετά σωστά από τους εισηγητές το θέμα της ε, ε, ελεύθερης έκφρασης της άποψης του καθενός για την πρόσβαση τώρα στα δημόσια έγγραφα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τον κανονισμό αυτό ως δικαιολογία για την μη πρόσβαση. Στο άτρο 7 τώρα. Μια έρευνα βάση μητρώων. αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και οι ιατρικές έρευνες. Γιατί έχουν ιδιαίτερη σημασία. Θεωρώ ότι θα είναι σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση σε κάποιες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα σήμερα να περιοριστώ σε θέματα οδηγίας, γιατί θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών μεταξύ των κρατών μελών. Για τη συνεργασία αυτή η οποία θα πρέπει να επεκταθεί, θεωρώ ότι χρειάζεται ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ε, εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών μελών. Και θεωρώ ότι χωρίς καμία αμφιβολία χρειάζεται και πιο καλή προστασία των δεδομένων. Αφενός αυτό είναι σημαντικό για την προστασία των ερευνών, αλλά και για την προστασία των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων και των μαρτύρων που συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες. Αναφέρεται σε κάποια κράτη-μέλη ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να αφορά μόνο διαευρωπαϊκές, συγγνώμη, διασυνοριακές υποθέσεις. Δεν συμφωνώ, γιατί πολλές φορές ξεκινούν σε εθνικό επίπεδο οι έρευνες και σε περτέρα στάδια μόνο αποκαλύπτονται διασυνοριακές διαστάσεις. Άρα είναι σημαντικό να υπάρχουν κάποια ελάχιστα πρότυπα σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων για να μην χρειαστεί εκ των υστέρων να διορθώνουμε καταστάσεις αλλά εξ αρχής να ισχύουν τα ίδια σε θέματα αστυνομικών ερευνών. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε σε τελική ανάλυση να υπάρχουν ίδια πρότυπα. Γιατί αν δεν το καταφέρουμε αυτό, δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Ευχαριστώ, κυρία Ρωμέρα Λόπες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους εισηγητέ για την προσπάθειά τους, ιδίως ε, για εναρμόνιση των δύο οδηγιών. Θα ήθελα όμως να μιλήσω για ένα ζήτημα το οποίο παράπλευρα μόνο το έχουμε θίξει μέχρι στιγμής, αλλά εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι πράγματι η οδηγία σε αυτές ε, ανταποκρίνονται στην πρόοδο τη τεχνολογίας που οδήγησε στην παγκοσμιοποίηση. Έχουμε λοιπόν αυτό το γενικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων που θέλουμε ε, να το ε, περικοδοτήσουμε με κάποια γενικά πρότυπα. Θέλω να σας πω όμως ένα παράδειγμα. Οι πολυεθνικές εταιρείε, οι οποίες ε, εγκαθίσταται σε διαφορετικέ χώρε. Α υποθέσουμε ότι επιβάλλονται κυρώσει σε κάποιες πολυεθνικές διεθνεί αυτέ τι μπορεί αυτέ να μην εντάσσονται σε αυτό το γενικό πλαίσιο. Όταν παραβιάζονται οι εγγύησεις στα ΕΧΕΓΕ και αυτό αφορά μόνο ένα εθνικό πλαίσιο. Όταν μιλάμε λοιπόν για γενικό πλαίσιο προστασία δεδομένων, δεν μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασία δεδομένων. Αυτό που λείπει είναι μια ευρωπαϊκή αρχή. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι στη συζήτηση να συμπεριλάβουμε το στοιχείο τη ανάγκη να υπάρξει και μια Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, η οποία θα καθορίζει ακριβώ ορισμένα κριτήρια, τα οποία μέχρι στιγμή ε, στο νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασία Δεδομένων δεν ορίζονται παρκώ. Διότι το Συμβούλιο έχει πολύ μικρέ και θα έλεγα και αδύναμε αρμοδιότητε και εξουσίε. Πολύ καλά είπε και ο κύριος Σάλβορ ότι δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο και η Κομισιόν δεν μπορεί να θεσπίσει αυτά τα τεχνικά πρότυπα. Γιατί δεν είναι αρμοδιότητα τη Κομισιόν, θα ήταν περισσότερο αρμοδιότητα αυτή τη Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασία Δεδομένων που δεν περιλαμβάνεται όμω στο πακέτο αυτό η συγκρότηση μια τέτοια αρχή. Θα πρέπει λοιπόν να το συμπεριλάβουμε στη συζήτηση και να δούμε πρέπει να προχωρήσουμε με τέτοια κατεύθυνση, να συγκροτήσουμε, να ιδρύσουμε μια τέτοια αρχή που θα θεσπίζει τα χέγγια, τις εγγυήσει. διότι βλέπουμε ότι σε εθνικό επίπεδο πολλέ φορέ ε, κατακλείζονται οι αρχέ από τέτοια φαινόμενα γενικά, παγκοσμιοποιημένα. Ο κύριος Κλοντ τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι στην ομάδα μα, αλλά και σε όλε. Ε, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα, το όλο ζήτημα. Το βλέπουμε και από τις αγωγικές παρεμβάσεις όλων των συναδέλφων. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, δύο εισηγητές ε, που έχουν καταρτήσει δύο πολύ καλές εκθέσεις. Ο πρόσωπος της Κομισιόν πολύ καλά είπε ότι μιλάμε και για προστασία των ατόμων αλλά και για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Άκρος πολύπλοκο λοιπόν το ζήτημα. Σίγουρα δεν θα μείνουν άπαντες ικανοποιημένοι. Για τη δική μας πολιτική ομάδα δύο είναι τα σημαντικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, όπως είπε και ο συνάδελφος ε, προηγουμένως από την ομάδα, θεωρούμε ότι και η οδηγία είναι πολύ σημαντική. Τα δύο μέσα λοιπόν, ο κανονισμός και η οδηγία θα πρέπει να ειδωθούν ως πακέτο και έχουμε μια γενική εξαίρεση προς τον γενικό κανόνα βέβαια με το διάλογο, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν αυτά τα δύο και σε ό,τι αφορά τη γλώσσα και του ορισμού και τι λοιπέ διατάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμά, ω πολιτική ομάδα. Και είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μα, παρότι πρόκειται για εισαγωγική συζήτηση, να ορίσουμε τουλάχιστον τι είναι σημαντικό για εμά ω ομάδε. Το profiling, χάρη, στο άρθρο 20, το ανέφερε ο συνάδελφο Δημήτρης Τρούτσας. Το άρθρο 20 είναι πάρα πολύ λεπτό ε, ο ζήτημα, αυτό το profiling δηλαδή. Και θέλουμε να επικεντρωθούμε σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει και οι ελεγκτέ δεδομένων που είναι κατεστημένοι εκτό Ένωση, αλλά παρέχουν υπηρεσίε ε, εντό Ένωση. Θα πρέπει να τους αφορά, θα πρέπει να καλύπτονται. Το έχουμε το ζήτημα της διαγραφής, το δικαίωμα να ξεχαστεί κάποιος. Ε, και πολλά άλλα ζητήματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και για ενδιαφερομένους φορείς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν με πνεύμα συνεργασίας να δουλέψουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σοσιαλδημοκράτε σίγουρα θα εργαστούμε σκληρά και θα συνεργαστούμε με όλους τους συναδέλφους για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν άρχισα να διαβάζω τις 217 αυτές σελίδες ε, πρέπει να πω ότι ελαφρώς ενοχλήθηκα κατά κάποιο τρόπο. Πρώτον, διότι ήταν λίγο αδύνατο ε, για τους ε, δύο εισηγητές, πιστεύω, να δεκπερώσαν τόσο ογκώδες έργο, αλλά και φιλοσοφικά, αν θέλετε, θέλω να κάνω σχόλιο. Η Κομισιόν ουσιαστικά τι έχει κάνει. Έχει ποντίσει ε, στη θάλασσα ένα ε, ημικατασκευασμένο, ημιναυπηγημένο πλοίο. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε την αυπήγηση, την κατασκευή. Και φοβούμαι ότι είναι λάθος. Είναι λάθος η κατασκευή κύριος Άλμπερχτ και ο άλλος ηγετής βέβαια, έχει ένα πρόβλημα που είναι λίγο αδύνατο να επιληθεί. Δηλαδή κάτι το οποίο από την αρχή έχει κατασκευαστεί λάθος, πώς μπορεί κανείς να το διορθώσει ή να το τελειοποιήσει. Πρώτα, ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στους υπόλοιπους ε, βουλευτές που θα ήθελα να λάβουν το λόγο. Πριν όμως στραφώ πάλι στους ηγητές, επειδή είμαστε πλέον επί Ιρλανδικής Προεδρίας, και η Ιρλανδική Πρόεδρε είναι αυτή η οποία θα πρέπει να αναλάβει την ε, πρόθεση αυτού του θέματος. Ε, έχουμε έναν εκπρόσωπο εδώ, τον κύριο Κόγκαν. Αν θέλει ο εκπρόσωπος της Ιρλανδικής Προεδρίας ε, να εκφραστεί, θα του δώσω τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε δεν επιμείναμε να ζητήσουμε το λόγο γιατί ξέρουμε ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος και ο υπουργό για τη Δικαιοσύνη και την Ισότητα ε, θα είναι την ε, θα είναι στην Επιτροπή σας κάποια στιγμή και θα τα πει ε, και σε εσά αναλυτικό, οπότε εγώ θα περιοριστώ σε κάποια γενικά σχόλια. Σίγουρα το ζήτημα είναι προτεραιότητα πάντως για την Ολλανδική Προεδρία και έχουμε ε, διαθέσει σημαντικούς πόρους στο να συνεχίσουμε την σημαντική αυτή προσπάθεια. Επίσης, Είχαμε πολύ καλές συναντήσεις με τους εισηγητές. Και βέβαια ασχολούμαστε πρώτα με τον κανονισμό. Η κυρία Ιντβελτ είπε πολύ σωστά ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε ε, γενικούς κανόνες πρώτα και μετά αναλυτικά να ασχοληθούμε με τις εξαιρέσεις. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε και θα συνεργαστούμε πολύ ευχάριστα μαζί σας και στους επόμενους έξι μήνες. Ευχαριστώ, λέω πρώτα στην Ελληνική Προεδρία. Ακούσαμε λοιπόν όλους τους βουλευτές και θα στραφώ τώρα στους δύο εισηγητές παρακαλώντας τους να ε, κάνουν μια συνθετική παρουσίαση των υπόψεων που άξουν. Πρώτα ο κύριος Άλμπρεχτ για τον κανονισμό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ συνάδελφοι για τα εκτενή σας σχόλια. Ασφαλώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και έτσι θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε ανοιχτά και εκκρεμή ζητήματα να σας πω ξεκάθαρα ότι βεβαίως και δεν είναι το τελευταίο σημείο αυτό το νομοθέτημα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση και το λέω αυτό γιατί αναγνωρίζω ότι κανείς σχεδόν δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Άρα πρέπει να τα συζητήσουμε εκτενώς και λεπτομερώς τα θέματα αυτά, αλλά κανείς δεν ξέρει πραγματικά ποια είναι η χρυσή λύση για κάποια τέτοια ζητήματα που αποσχολούν την κοινωνία. Είμαστε όμως στο σωστό δρόμο. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα τις εργασίες μας και πολλές από τις αλλαγές που έγιναν που προτάθηκαν βασίστηκαν στις συζητήσεις που έχουμε ήδη κάνει. Ασφαλώς και θα είμαι ανεκτός για συμβαστικές προτάσεις σε ό,τι αφορά και τις τροπολογίες που έχουν καταδεθεί. Να πω τέλος ότι θεωρώ ότι η οικονομική ανάπτυξη και η προστασία των δεδομένων δεν αποτελούν διφαντικούς όρους και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να τονίζουμε ξανά και ξανά. Τι κάνουμε εδώ, προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των πληροφοριών μεταξύ των δύο μερών που συμφωνούν για την συναλλαγή μεταξύ των ε, πελατών και των επιχειρήσεων ουσιαστικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν ο κόσμος θέλει να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία να μπορεί να το κάνει βάσει κάποιων κανόνων. Αρκεί να, έχουν, να έχει και στην διάθεσή του τα στοιχεία που χρειάζεται. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, θεωρώ ότι αυτές θα ωφεληθούν ιδιαίτερως, γιατί ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μικρών και των μεγάλων επιχειρήσεων οι καταναλωτές, οι πολίτες είναι το πιο αδύναμο μέρος. Δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν πλήρως και να υποφεληθούν πλήρως από τον ανταγωνισμό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας αλλά και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού θεωρώ ότι τα πρότυπα και οι κανόνες προστασίας δεδομένων σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών, των καταναλωτών. Αυτό είναι καθοριστικό, ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον, αλλά και παντού. Γιατί φυσικά υπάρχει μεγάλη διασύνδεση σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε πλέον το ψηφιακό από το αναλογικό περιβάλλον. Στο πνεύμα λοιπόν αυτό σας καλώ να μας βοηθήσετε να πετύχουμε αυτό το στόχο που πολλές φορές έχει αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και με μεγάλη μου χαρό, χαρά να διαθέσω όλο το χρόνο που διαθέτω σε συνεργασία με την Ιρλανδική Προεδρία προκειμένου να πετύχουμε, ελπίζω, το στόχο μας. Προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πριν από τις ευρωεκλογέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Άλμπρεχτ και τώρα κύριε Τρούτσα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. Ε, έχουμε τηρήσει το χρονοδιάγραμμά μα. Θα ευχαριστήσω λοιπόν όλου του συναδέλφους για τι συμβολέ του, τα καλά του λόγια και την, ε, τα ενθαρρυντικά τους λόγια, αλλά και για τις πιο επιφυλακτικές παρατηρήσεις και για τις προτάσεις που ήδη έγιναν. Αυτό δείχνει σαφώς πόσο σημαντική είναι αυτή η υπόθεση της μεταρρύθμισης της προστασίας των δεδομένων και ε, συμφωνούμε ότι είναι τεράστια σημασία για τους συμπολίτες μας και γι' αυτό και εκτιμώ τα σχόλια του Προέδρου ότι θα δοθεί περισσότερο χρόνο στην Επιτροπή μας για περισσότερη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος. είναι σαφές και λογικό να δίνετε τόση προσοχή σε αυτόν τον ε, κανονισμό και όχι στην οδηγία. Είμαι ρεαλιστής και πάνω σε αυτό το θέμα. Συμφωνώ επίσης με τα όσα είπε η Σόφη Ιντεβέλντ ότι αυτή η οδηγία θα πρέπει να θεωρηθεί ως εξαίρεση γιατί ακολουθούν και άλλα θέματα. Ο κανονισμός είναι το βασικό κομμάτι της δουλειάς μας. Αλλά να επαναλάβω και να τονίσω άλλη μια φορά ότι η ουσία που θα πρέπει να συζητήσουμε σε σχέση με την οδηγία της επόμενης εβδομάδας και μήνες είναι το πολιτικό θέμα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με αυτή την οδηγία και που θα εξαρτηθεί από το πώς το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη θα αντιδράσουν, πώς θα συνεχίσουν τη δουλειά για το θέμα αυτό. Μπορεί δηλαδή και το Κοινοβούλιο να χρειαστεί να αντιμετωπίσει από πολιτικής άποψης αυτό το θέμα. Ευχαριστώ και πάλι όλους. Και εμείς σας ευχαριστούμε τους εισηγητές και το μέλη που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση που ήταν ε, εις βάθος, αλλά μπορούμε να κάνουμε και άλλη μία σε δύο εβδομάδες ε, ε, από τώρα δηλαδή 2021, σε δύο εβδομάδες που έχουμε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής μας και μπορούμε να δώσουμε μια δεύτερη συζήτηση τότε, να κάνουμε μάλλον μια δεύτερη συζήτηση τότε. Ε, προθεσμία ε, για κατάθεση τροπολογιών 27 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Είναι ε, συνήθιστα μακρύ το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή τροπολογιών. Έτσι ώστε να έχουμε χώρο να ελέγξουμε και να δούμε πώς θα προχωρήσει η συζήτηση. Πώς πάει μάλλον η συζήτηση για να διατηρήσουμε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Άλβαρο, θέλετε κάτι να πείτε. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή περίμενα να αναφέρετε την προθεσμία για υποβολή τροπολογιών. Σε σχέση με τις συνήθεις προθεσμίες που έχουμε, είναι ήδη μακρά. Τώρα βέβαια μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το κατά πόσο αρκεί η συνήθιση σε προθεσμία που έχουμε μια-δύο εβδομάδες δηλαδή. Τώρα στην περιπλοκότητα του θέματος και την αλληλεξάρτηση της οδηγίας και του κανονισμού, την αλληλοσύ... τη σύνδεση μάλλον και τα πολλά σαφήνιστα ερωτήματα και έχοντας υπόψη ότι ένα έτος προετοιμαζόταν ε, οι επιτροπές, οι σκιώδεις ε, δούλευαν πάνω σε αυτό και άρα ε, η συμβολή των εισηγητών είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα να ζητήσω αν είναι δυνατόν να εξετάσουμε τη δυνατότητα μετακίνησης της προθεσμίας στα τέλη Μαρτίου αντί για τα τέλη Φεβρουαρίου γιατί να αποφασίσουμε κάτι είτε από την άποψη επιβολή νόμου, είτε από την άποψη ισορροπία μεταξύ οικονομικών συμφερόντων και καταναλωτών. Επηρεάζονται 500 εκατομμύρια άνθρωποι. Ε, δεν θα ήθελα να λάβουμε βιαστικέ αποφάσει πριν να μπορέσουμε να μελετήσουμε ει βάθο το θέμα. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα και όχι στο χρόνο. Και νομίζω πως μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες των εισηγητών και να γίνει η ψηφοφορία υπό την Ιρλανδική Προεδρία. Ναι, έγινε μια πρόταση. Δεν ξέρω πώς αλλιώς παρά να παραπέμψω το θέμα στους εισηγητές και τους κοιόδης εισηγητές να το συζητήσουν εκείνοι. Δεν ξέρω, με γραπτή διαδικασία μέσα στις επόμενες ώρες πρέπει να ληφθεί απόφαση τώρα. Γιατί έχουμε δεύτερο γύρο για τη συζήτηση σε δύο εβδομάδες. Ίσως θα μπορούσαν να, να μεταξύ να το συζητήσουν, να συζητήσουν και με τους σκιώδεις και να δούνε αν αυτή η ασυνήθιστα μακρά διαδικασία υποβολή τροπολογιών θα πρέπει να παραταθεί για κάπου στο Μάρτιο. Άρα λοιπόν καλό είναι να, οι εισηγητές να κάνουν, ε, να, το αποφασίσουν μαζί με τους σκιώδεις. Άλμπρεχτ. Ναι, ε, να αναφερθώ μόνο σε αυτό και να πω ότι ήδη έχουμε κάποια ανταλλαγή απόψεων για την ε, προθεσμία τροπολογιών. Ο συγκητή και οι σκιώδες είχαν, συμφωνήσει για αυτή την προθεσμία 27 Φεβρουαρίου και όπως είπε ο κύριος Άλβαρο ήδη είναι μακρά η, προθεσμία και θα είναι δυνατόν να ανασταλούν τροπολογίες μέχρι τον Φεβρουάριο. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να βρούμε συμβιβαστικέ. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα πάρουμε χιλιάδες ε, τροπολογίες και το πρόβλημα θα είναι πώς μετά θα ψηφίσουμε. για να μπορούμε να διαπραγματευτούμε και με την ελληνική Προεδρία. Ο Δημήτρης Δρούτσε. Εγώ συμφωνώ με τα όσα είπε ο Γιάνν Άλμπρεχτ. Εγώ ευχαρίστω να είμαι ευέλικτο, Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ισορροπήσουμε. Ξέρουμε τα επιχειρήματα, ξέρουμε το άγχος όλων, αλλά πρέπει να μείνουμε σε μια ισορροπία την οποία ήδη έχουμε φτάσει, κατά τη γνώμη μου είναι κάπως πρόημο να αποφασίσουμε για παράταση της προθεσμίας σε αυτή τη φάση. Όμως θα ήθελα εγώ μια διευκρίνηση από την Ιρλανδική Προεδρία, γιατί είπατε ε, κάτι που με μέρδεψε. Είπατε ότι το Συμβούλιο σκοπεύει να κάνει μια διοχική συζήτηση για τον κανονισμό και την οδηγία. Και τώρα που μιλάμε για χρονοδιάγραμμα, εμείς επιμένουμε για την προσέγγιση πακέτου και μάλιστα η οδηγία είναι μια προϋπόθεση για την υιοθέτηση άλλων θεμάτων άλλων ντοσιέ με τα οποία ασχολείται το Συμβούλιο για τη... στον τομέα της αστυνομική και δικαστικής συνεργασίας. Θα ήθελα λοιπόν να έχω μια εξασφάλιση ε, από το Συμβούλιο ότι ταυτόχρονα και παράλληλα θα δουλέψετε για αυτήν την οδηγία και όχι διαδοχικά η Ιρλανδική Προεδρία. Ξέρω πως έχουμε λίγο χρόνο. Ευχαρίστως θα μπορούσα να μιλήσω με την κυρία Εντβέλτ. Εγώ δεν είπα ότι θα γίνει διαδοχικά. Είναι κοινή προσέγγιση στο πακέτο. Απλώς είπα ότι θα ασχοληθούμε πρώτα με τον κανονισμό, γιατί όπως είπατε χρειαζόμαστε ένα γενικό κανόνα πριν να συζητήσουμε ε, τις λεπτομέρειες και τις εξαιρέσεις. Οι συνάδελφοι της προηγούμενης Προεδρίας ανακάλυψαν ότι υπήρχαν πολλές επαναλήψεις στη συζήτηση όταν προσπάθησαν να γίνουν οι συζητήσεις αυτές παράλληλα. Όλα λοιπόν αυτά θα γίνουν από την Ιρλανδική Προεδρία. Απλώς σκοπεύαμε να ασχοληθούμε πρώτα με τον κανονισμό. Ο κύριος Φως, ευχαριστώ πολύ. Φυσικά πολύ ελκυστικό είναι να γίνει αυτή η αναβολή γιατί πολλά θέματα και πολλά προβλήματα θα το προαπαιτούσαν αυτό. Αλλά φυσικά στην παρούσα φάση αντιμετωπίζουμε και μια χρονική πίεση και θα πρέπει να τα αποκριθούμε. Θα, θέλαμε, θα ήθελα λοιπόν η απόφαση για την τήρηση ή μη της προθεσμίας να ληφθεί κάποια στιγμή αρχές Φεβρουαρίου. Να δούμε αν μας φτάνει ο χρόνος ή όχι. Για να εργαστούμε πιο συγκεντρωμένα και να πάρουμε στην πορεία την απόφαση κατά πόσον θα χρειαστεί ή όχι αναβολή. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, νομίζω ότι καταλήγουμε σιγά σιγά σε μια συμφωνία, θα τηρήσουμε επί του παρόντος το χρονοδιάγραμμα και θα γίνει μια δεύτερη συζήτηση σε δύο εβδομάδες. Θα δούμε πώ θα πάνε τα πράγματα μέχρι τότε. Νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η πρόταση και ισορροπημένη. σε ό,τι αφορά και την ε, προθεσμία για την υποβολή ε, τροπολογιών. Σε δύο σχεδόν μήνες, μάλιστα. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω στην ημερήσια διάταξη, αλλά έχουμε ακόμα μία ευκαιρία να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας, εάν ε, είμαστε γρήγοροι στο επόμενο πακέτο. Please. Those of you leaving the room. Παρακαλώ. Όποιοι φεύγετε, ησύχω παρακαλώ. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε εμείς με την ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ. Αναλαμβάνω, μην κάνετε θόρυβο βγαίνοντα από την αίθουσα για να μπορέσουμε εμείς να προχωρήσουμε γρήγορα. Όπως σας είπα, έχουμε τώρα μια κοινή συζήτηση διαπερισμένων ζητημάτων των σημείων 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15. Όλα αυτά τα σημεία αφορούν την απαλλαγή για το 2011 διάφορα τμήματα του Γενικού Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Το τμήμα 3 Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Ελεγκτή Προστασία των Δεδομένων, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, τη Eurojust, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία ΣΥΠΟΛ, τον Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ένωσης, τη Frontex δηλαδή, τον Frontex μάλλον, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία Europol και τέλος ε, επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχο των οργανισμών. Όλα αυτά τα θέματα τα έχει εξετάσει ένας και μόνος εισηγητής, ο συνάδελφός μας Γιώργος Παπα-Νικολάου, Προτείνω λοιπόν να ακούσουμε συνοπτικά την παρουσίαση των σχεδίων γνωμοδότησης για την απαλλαγή για τα σημεία που προανέφερα από το 7 έως και το 15 και συνεχεία θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δώσουμε το λόγο και σε κάποιον εκπρόσωπο της Κομισιόν ή σε άλλους συναδέλφους βουλευτές. Κύριε Παπα-Νικολάου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πραγματικά σύντομος γιατί ξέρω ότι πολύ λίγος χρόνος έχει μείνει. Μιλάμε για την τελική έγκριση λοιπόν ε, του προϋπολογισμού μετά την ολοκλήρωση των ελεγμένων λογαριασμών με βάση τη συνθήκη και τους κανόνες μας πρέπει να εγκριθούν και από, τον, ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαδικασία απαλλαγή ουσιαστικά θα εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο οι Κομισιόν και οι οργανισμοί που αναφέρατε εφάρμοσαν τον προπολογισμό του για το 2011 και πώ έκλεισαν οι λογαριασμοί του βασιστήκαμε σε κάποιες εκθέσεις και το Ελληνικού Συνεδρίου, την ε, δήλωση αξιοπιστίας και τις απαντήσεις που έδωσαν οι οργανισμοί και τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Μιλάμε για τον εξωτερικό έλεγχο, που επίσης ε, είναι κάτι σημαντικό για εμάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή Κοντ βέβαια, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Έλεγχου είναι ε, υπεύθυνη. Εμεί γνωμοδοτούμε για του οργανισμού που εμπίπτουν στον τομέα τη ελευθερία δικαιοσύνη και ασφάλεια και στο σχετικό τμήμα της, ε, που αφορά την Κομισιόν του 3 δηλαδή. Εμεί, λοιπόν θα συντάξουμε σχέδια γνωμοδότηση για την Επιτροπή λοιπόν ε, Ελέγχου του Προπολογισμού και για την Επιτροπή, το Τμήμα 3 και για τις διάφορες από τους οργανισμούς στους οποίους αναφέρατε που επίπτουν στον τομέα ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας. Επίσης έχουμε και μια γενικότερη γνωμοδότηση για τις επιδόσεις δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχο των ε, οργανισμών. Βασιζόμαστε στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και στα σχόλια των οργανισμών για την έκθεση του ελεκτικού. Έχουμε δει επίσης και κάποια άλλα στοιχεία για να δούμε αν ήταν θετικές ή αρνητικές οι πρακτικές στους τομείς δικαιοσύνης, εσωτερικών και κτλ. Τώρα, πιο συγκεκριμένα και με βάση τις πληροφορίες που έχουμε λάβει, για αυτούς τους οργανισμούς που προανέφερα, Βλέπουμε ότι υπήρξαν πολύ σωστές τακτικές, κανονικές νόμες διαδικασίες, δεν είχαμε μεταφορά ε, σημαντική Ε, σωστές από τις 7, Σέπολ, Euro, Just Frontex. Υπάρχει εξήγηση βέβαια για το ότι εν μέρει εξαρτάται και από κάποιες εξωτερικούς παράγοντες ε, η εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών αυτών. Για τη Frontex πριν από κάποιες εβδομάδες είδαμε ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα. Also. In the case of Frontex in particular, the agency received uh, funds worth 31.8 million in late October 2011. Additional funds Μιλάμε για κάποια επιπλέον ποσά της Τάξη 31,5 ε, και τα έχουμε αναφέρει και στην ομοδότησή μας. Και προάλλα προβλήματα είχαμε και υπάρχουν και τομεί που μπορούμε να έχουμε βελτίωση. Το λέει και το ελεγκτικό συνέδριο. Και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ε, διαχείριση. Η ΣΕΠΟΛ έχει βελτιωθεί σε ό,τι αφορά το 2008 που δεν είχε πάρει απαλλαγή. Βέβαια πολλά ακόμη θα πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση αδυναμιών στον προγραμματισμό. Πάντως ε, είναι στο σωστό δρόμο οι οργανισμοί. Κάτι άλλο που μας ανησυχεί είναι κατά πόσον μπορεί η αστυνομία, η αστυνομική ακαδημία να συνεχίσει να ε, στεγάζεται στο κτίριο, στον πράξη ρόλοι ευθύνε μεταξύ ε, του διευθυντή και των υπόλοιπων μιλών του Eurojust είναι ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί και για το Γιούρτζα να πω κάτι ακόμη για την απαλλαγή. Η πρότασή μας και η πρόθεσή μας είναι στην επόμενη θεώρηση του κανονισμού Γιούρτζα να δούμε πιο λεπτομεριακά αυτά τα θέματα. Σε ό,τι αφορά τον οργανισμό, το κέντρο μάλλον Παγκοσμίου το Τοξικομανία, είχαμε κάποιο ποσοστό τάξη των 270.000. Δεν βρήκαμε μία λύση. Δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό το ποσό και είχαμε και το ζήτημα της μίσθωσης ε, των ε, γραφείων που θα πρέπει ή να ενοικιαστούν ε, ή να απολυθούν και πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό. Και είναι δύσκολο μέσα σε κρίση. Τέλο, για τον και των δικαιωμάτων, και δεν έχουμε κανένα σημαντικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα ακόμη που θα ήθελα να σας αναφέρω και κλείνω. In, in our auditing for the future, the, the, the court of auditors... Όπως προκύπτει και από τους εξωτερικούς ελέγχους και από το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση ε, στον έλεγχο των επιδόσεων για να είμαστε βέβαιοι ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δαπανώνται με ορθολογικό τρόπο. Έχουμε μια δημοσιονομική κρίση, περίοδο λιτότητα διανύουμε, άρα οι οργανισμοί τη Ένωση θα πρέπει να δαπανούν με σοφό και αποτελεσματικό τρόπο τα χρήματα που του διατίθενται. Θέλω να ευχαριστήσω τέλο τη γραμματεία μα, ε, την κυρία Κατρίν Χιούμπερ, για την πολύ καλή συνεργασία που είχα μαζί της κατά την κατάρτιση των εκθέσεων. Αυτό σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και εσάς κύριε Πρόεδρε. Προσπάθησα τα πω όλα πάρα πολύ σύντομα. Summarized. Σας ευχαριστούμε κύριε Παπα-Νικολάου για την παρουσίαση αυτή τη συνοπτική όλων των σχεδίων έκθεσης σε ό,τι αφορά την απαλλαγή προκειμένου να ολοκληρώσουμε ε, γρήγορα. Και έτσι έχουμε κάποιο χρόνο να ακούσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια σχόλια. Έχουμε μαζί μας κάποιον εκπρόσωπο της ευρωπαϊκή επιτροπή; Μάλιστα, την κυρία Μακοβάη. Έχετε το λόγο. Thank you for giving me the floor. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστήσω και τον εισηγητή του κ. Παπα-Νικολάου για την ισορροπημένη αυτή έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάποιο σχόλιο για το σχέδιο της έκθεσης. Θα θέλαμε μόνο να παρουσιάσουμε την θέση μας σε ό,τι αφορά την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο που μας αφορά και να αναφέρουμε και κάποιες γενικές παρατηρήσεις για τα θέματα αυτά που αναφέρονται στην έκθεση για το κεφάλαιο 8. Για το κεφάλαιο 8 του ελεγκτικού συνεδρίου χαιρόμαστε, το καλωσορίζουμε, χαιρόμαστε που δεν εντοπίστηκαν ατασταλίες και αυτό σημαίνει ότι τηρήσαμε τις ε, οικονομικές διατάξεις. Τώρα για τα θέματα που αναφέρονται στο σχέδιο έκθεσης σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προτάσεις του εισηγητή. Για το πρώτο θέμα σε ό,τι αφορά την έλλειψη πληροφοριών σε ό,τι αφορά την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Αυτό ασφαλώς αποτελεί αρμοδιότητα του ελεκτικού συνεδρίου. Αυτό αποφασίζει τη μεθοδολογία που ακολουθεί για το θέμα του αυξημένου επίπεδου εφαρμογών σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις και τις πληρωμές για το 2011 διαπιστώνουμε ότι και για το 2012 τα προκαταρτικά στοιχεία καταδεικνύουν υψηλό επίπεδο πληρωμών και δεσμεύσεων. Για το τρίτο θέμα, για το κεφάλαιο 1807, 02, συγγνώμη, μπορούμε να πούμε με ικανοποίηση ότι και αυτή η εφαρμογή ήταν πάρα πολύ καλή, 97% επίπεδο, που σημαίνει ότι ήταν καλό το επίπεδο δημοσιονομικού προγραμματισμού σε ό,τι αφορά την ετήσια έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης ε, Ιστορικών Υποθέσεων για το 2011, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι ακολουθήσαμε όλα τα μέτρα τα οποία είχαμε προαναγγείλει και σε ό,τι αφορά την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητε του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει εκτενώς τα αποτελέσματα για να γίνει και σχετική αξιολόγηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να ακούσουμε μήπως κάποιοι βουλευτές θα ήθελαν να πάρουν το λόγο. Κυρία Ματιό, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο για τις εξαιρετικές εκθέσεις, για αυτές ε, τις πολύ σημαντικές ε, απαλλαγές και μάλιστα ήταν πολύ σημαντικό να τις δούμε αφού τελείωσε το προηγούμενο θέμα γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι αυτοί οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που μας αφορούν εδώ στη ΛΥΜΠΕ είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και είναι κρίμα που δεν ενδιαφέρει περισσότερους στην αίθουσα. Αλλά, εν περιπτώσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Για να έρθουμε στα δικά μας. Οι οργανισμοί μας απασχολούν σήμερα είναι πολύ σημαντική και είμαστε ικανοποιημένοι γιατί το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο δεν έχει εκφράσει καμιά επιφύλαξη για την ε, δημοσιονομική διαχείριση των οργανισμών. Όμως, ε, και το είπε και ο συνάδελφο, είναι αλήθεια πως το Ελεκτικό Συνέδριο όλο και λιγότερο ε, περιλαμβάνει τέτοιες φράσεις και περιορίζονται οι εκθέσεις, σμικρίνονται κάθε χρόνο και μικρότερες ε, οι εκθέσεις και μάλιστα η έκθεση που είδαμε για τον Οργανισμό δικαι... Ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι πολύ πολύ μικρή. Ενώ κάθε χρόνο εκδίδονται γνωμοδοτήσεις ε, και διαμαρτυρόμαστε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, αλλά δεν γίνεται τίποτα δυστυχώ. Να πω δύο λόγια για την ΣΕΠΟΛ. Είναι αλήθεια ότι το 10 αρνηθήκαμε την απαλλαγή στην ΣΕΠΟΛ, γιατί υπήρχαν πολύ σημαντικά προβλήματα με τον προηγούμενο διευθυντή. Αλλά ήθελα να αναφέρω και το έχουμε πει κάθε φορά, ότι ο σημερινό διευθυντή έχει κάνει πολύ σημαντικές προσπάθειες και ότι η διαχείριση είναι αυτή τη στιγμή τέλεια. Έχει μειώσει το κόστος το λειτουργικό έχει κάνει κάποιες μετακινήσεις του προσωπικού εκεί που έπρεπε και η διαχείριση αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά τέλεια. Και όσον αφορά το Eurojust, το είπε και ο συνάδελφος ότι εκεί ίσως ε, δώσαμε στον διευθυντή νομική βάση λανθασμένη και θα πρέπει να τη διορθώσουμε φέτος. Αλλά εν γέννη, οι γενικοί διευθυντές είναι στην ουσία από διοπομπαίος στράγος κάθε φορά. Ε, τους, βάζουμε, τους τα ρίχνουμε όλα αυτονών αλλά γενικά πρέπει να δούμε και τις νομικές βάσεις ε, και είχα ζητήσει σε κάποια φάση στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού ε, να ορίσουμε έναν υπάλληλο του Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα, αντιπροσωπεύεται, θα εκπροσωπείται με ε, συμβουλευτική ψήφο και συμμετοχική ψήφο και έτσι αποφεύγουμε διάφορα λάθη. Όπω είδαμε στις ΕΠΟΛΑ, α πούμε. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο τότε, Θα είχαμε αποφύγει τα προβλήματα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, είχα να πω και ευχαριστώ και πάλι για το δουλειά που έκανες. Ευχαριστούμε κυρία Ματιέ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο για αυτό το σημείο. Αν όχι, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπα-Νικολάου. Σας ευχαριστούμε για... και για την ε, συνοπτική εκδοχή και την παρουσίαση της... του σχεδίου έκθεσης, γιατί έτσι θα έχουμε χώρο, χρόνο για να ανακοινώσουμε ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών έχει οριστεί στις 21 ε, Ιανουαρίου. 21 Ιανουαρίου το μεσημέρι. Στις 12, εντάξει. Το έχετε σημειώσει όλοι. Οπότε μόλις ε, έχουμε το χρόνο για να προετοιμαστούμε για τις εξής ψηφοφορίες. Τι είναι εξής ψηφοφορία. Η ψηφοφορία για τα σχέδια γνωμοδότηση θα πρέπει να γίνει στα τέλη, στα τέλη Φεβρουαρίου 2021. Τις, ε, τα σχέδια χνομοδότησης που παρουσίασε ο συνάδελφος Παπα-Νικολάου δηλαδή. Τώρα, δύο σημεία της μερικής διάταξης έχουν αναβληθεί και θα πρέπει να προχωρήσουμε. For the vote in minutes. minutes from... Σε δύο λεπτά ξεκινάμε τις ψηφοφορίες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

just when we got started this morning, I said two things. First first. Happy New Year. Λοιπόν, τα είπα και το πρωί, αλλά πριν αρχίσουμε τις προφορίες θα τα ξαναπώ. Καλή χρονιά σε όλους για όσους δεν ήταν εδώ το πρωί. Δεύτερο, να πω ότι θα πρέπει να έχετε την ηλεκτρονική σας κάρτα ψηφοφορίας. Στείλτε κάποιον να σας τη φέρει. Βλέπω πως κάποιοι συμμετέχουν μεν στην ψηφοφορία, αλλά δεν έχουν την ηλεκτρονική του κάρτα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώ δεν θα είναι πολύ μακριά η ψηφοφορία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν λοιπόν κάποιο έχει το δικαίωμα να ψηφίσει, αλλά δεν έχει την κάρτα του... Electronic Σας παρακαλώ απλώς να μου το πείτε ώστε να σας μετράμε. We can account for the members who do not have the να μετράμε όσους δεν έχουν την κάρτα τους. Τέσσερις άκαρτοι. Πω δεν θα είναι εύκολο <laughs> να σας μετρήσουμε. Λοιπόν, μόνο ένα θέμα έχουμε. Και ο εισηγητής είναι ο κύριος Φίλιπ Κλέης, που δεν έχει την κάρτα του από πάνω. So please make sure that your vote is taken into account. Λοιπόν, Κάθε φορά λοιπόν να μας λέτε τι ψηφίσατε. Σχέδιο γνωμοδότησης λοιπόν. Please, Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ησυχάστε και συγκεντρωθείτε. Τι έχουμε εδώ, τι μετανάστευτο των μεταναστών. Οι επιπτώσεις ε, στην αγορά εργασία, στην κοινωνική, στην, στην κοινωνική ασφάλιση κτλ. Ο συγκεκριτή είναι ο κ. Φίλιπ Κλέη. Θέλετε να σχολιάσετε. Όχι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία αυτή τη έκθεση. Ως έχει και βρίσκεται. Ξεκινάμε λοιπόν. Αν είστε όλοι έτοιμοι, τροπολογία 1 υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Those against. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 6 έχει αποσυρθεί, 5 έχει καταπέσει, 4 έχει παρακαταπέσει, 7 υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο τώρα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά αντροπολογία 9. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος. 11 κατά 31 απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 και 20 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, ελέγχουμε 13 και 20 ελέγχουμε τέλος ψηφοφορίας 26 κατά 18. Ε, έναντι 18. Εγκρίνεται. 20 και 21 μαζί. Ε, που είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά... Α, με συγχωρείτε. 21 και 22 είναι που ψηφίζουμε μαζί, γιατί είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνονται. 24 και 26. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνονται 27 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 27 άρχεται ο έλεγχος η ψηφοφορία μάλλον τέλος 19 28 απορρίπτεται 29 favor. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Α, όχι. Συγγνώμη. Έχει καταπέσει. 30 έχει καταπέσει. 31 έχει καταπέσει. 32 έχει καταπέσει. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35. Όχι, συγγνώμη, εγκρίνεται, εγκρίνεται, ναι. Το είπα λάθος, αλλά ας το ελέγξουμε. 34, άρχεται η ψηφοφορία, 34. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ναι, έκανα λάθος. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 πέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 και 38. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 41 και 42 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ να ελέγξουμε για τη 46 ελέγχουμε για τη 46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 Δεδομένων των τροπολογιών που εγκρίθηκαν και θεωρώ ότι ριζικά αλλάζουν τη φιλοσοφία του κειμένου, θα ψηφίσω κατά. Θα καταψηφίσω αυτή την έκθεση και σας συστήνω το να κάνετε το ίδιο. Και αν εγκριθεί θα ήθελα το όνομά μου να διαγραφεί από την γνωμοδότηση αυτή. 27 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται και σημειώνουμε και ότι θέλετε να διαγραφεί το όνομά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κλάς για την δουλειά που έκανε. We should be moving. We Μάλιστα, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε στις ψηφοφορίες. Και πάλι, σας παρακαλώ να φύγετε χωρίς πασαρία, για να μπορέσουμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Στο 18 περνάμε. Για την δέσμευση και δίμευση των προϊόντων του εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μακοβέη είναι η συγγήτρια. Αν θα θέλετε παρακαλώ να αποχωρήσετε ησύχως. Μισό λεπτό κυρία Μακοβέη, μισό λεπτό αν θέλετε για να υπενθυμίσω σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα σχετικό θέμα για τη δέσμευση και τη δίμευση των προϊόντων του εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση οδηγίας παρουσιάστηκε το 2012 και ο σκοπό έχει να μεταρρυθμίσει το νομικό πλαίσιο για τη δέσμευση και τη δίμευση σε περίπτωση ενδεχόμενου κινδύνου το σχέδιο της έκθεσης Το παρουσίασε η κυρία Μακοβέη, η συγγήτρια, στις 19 Σεπτεμβρίου του 2012. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είχε οριστεί στις 13 Δεκεμβρίου. Εν τω μεταξύ το Συμβούλιο βρήκε μια κοινή προσέγγιση για το κείμενο. Θα μας μιλήσει η κυρία Μακοβέη για το πώς έχει κατάσταση σήμερα. Έχετε τώρα το λόγο κυρία Μακοβέη. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω του συναδέλφου για το ενδιαφέρον που δείχνουν ε, για το θέμα αυτό. Θέλω να του ευχαριστήσω και για τι τροπολογίε του. Προσωπικά μαζί με του κοιόδου συζητητέ, Προσελίνο Αλφάνο, καταθέσαμε τροπολογίες για να ενισχύσουμε τις διατάξεις που αφορούν ε, την ε, δίμευση που δεν, κατα, ε, που δεν βασίζεται σε καταδίκη και κάποιες άλλες περιπτώσεις κατασχέσεων δημεύσεων για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα, ιδίω ό,τι αφορά και τις απαιτήσει για δίκη δίκη. Πρόκειται για τροπολογίες οι οποίες έχουν στόχο πρώτον την Διευκρίνησε ότι η δίμευση, η κατάσχεση μπορεί να διαταχθεί μόνο από τις δικαστικές αρχές. Δεύτερον, να διευκρινίζουν ότι οι μη ε, μάλλον οι δήμες που δεν βασίζονται σε καταδίκη μπορούν να διατάσσονται μόνο όταν το δικαστήριο δυνάμει των περιστάσεων των ειδικών μιας υπόθεσης θεωρήσει ότι ουσιαστικά ε, πρόκειται για περιουσία που αποκτήθηκε από παράνομη εγκληματική δραστηριότητα. Επίση, πρέπει να υπάρχουν σαφεί διατάξει για το σεβασμό του δικαιώματο υπεράσπιση ε, του δικαζόμενου και επίση την αρχή τη καλή πίστη των τρίτων μερών. Επίση, υπάρχει ανάγκη τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν νομοθετικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν ε, την πρακτική ε, πλασματικής μεταβίβασης της περιουσίας σε τρίτους για να μην υπάρξει πάγωμα ή κατάσχεση της περιουσίας. Πέμπτη κατηγορία. Πρέπει να ενισχυθεί το ότι η θυγόμενη από την απόφαση περιδίμευσης ή κατάσχεση θα πρέπει ή να έχουν ε, την συνδρομή δικηγόρου σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και έκτον η κατασχεθήσα περιουσία θα πρέπει κυρίως να χρησιμοποιείται για σχέδια πρόληψης εγκλημάτων ή άλλα σχέδια που είναι ε, προς το κοινό συμφέρον. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που κατέθεσαν τροπολογίες. Οι τροπολογίες αυτές αφορούν κυρίως κάποιες εξαιρέσεις όπου δεν θα πρέπει να υπάρχει όχι αυτή η διάταξη όταν είναι δυσανάλογο το βάρος που επιβάλλεται στο άτομο ή μπορεί να μην μπορεί να υποστηριχθεί κάποια αξίωση, κάποιο χειρισμό ε, του θύματος κατά του δράστη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα και την επέκταση ε, της ε, δίμευσης και σε αυτούς, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τα διαθέσιμα για τη λήψη μιας σχετικής απόφασης. Και υπάρχουν και πολλέ τροπολογίε που προβλέπουν τη διαχείριση και κοινωνική επανάχρηση της δημευθύσας σα περιουσία για να μην χαθεί αξία της και βέβαια για να μην έχουμε και περαιτέρω δηματική διείσδυση. Ε, συντομία αυτές είναι οι κύριε ομάδε των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί και οι υπόλοιποι σκιώδεις και εγώ Νομίζω ότι έχουμε ακολουθήσει κατά βάση μια γενική προσέγγιση για την έκθεση αυτή. Αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι η οδηγία για τις κατασχέσεις και δημεύσεις να είναι ισχυρή. Να περιλαμβάνει τις δημεύσεις τριτών μερών, εκτεταμένη δήμευση, δήμευση που δεν βασίζει κατά δύο κτλ. Ελπίζουμε να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία όπως και προηγουμένως όταν μάλλον όπως και μέχρι τώρα όσο, όποτε έχουμε συζητήσει την ε, πρόταση αυτή. Να πω επίσης ότι κατόπιν αιτήματος πολιτικής ομάδας η ψηφοφορία στην Επιτροπή να βάλετε για την 21η Ιανουαρίου. Συγγνώμη, διορθώνω, 31η Ιανουαρίου. Και τώρα περιμένω ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μακοβέη. σκιώδης τώρα. Με ποιον να ξεκινήσουμε. Ρίτα Μπροσελίνου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, πριν από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που όπως και εγώ είναι μέλος ε, της Επιτροπής ΚΡΙΜ και ξέρει πόσο σημαντικό είναι να φτάσει σε καλό συμπέρασμα. Ξέρουμε σε επαφές που είχαμε με τις αστυνομικές αρχές, με εκπροσώπους των πολιτών στις διάφορες ακροάσεις που είχαμε. Το να πλήξουμε το οργανωμένο έγκλημα μέσω της κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων σημαίνει ε, να περιορίσουμε, να εμποδίσουμε βασικά. Η Κομισιόν ε, μας έκανε μια πρόταση που θα έλεγα εγώ πως είναι κάπως επιφυλακτική. Εμείς πρέπει ως Ευρωκοινοβούλιο να το ενισχύσουμε και να το καταστήσουμε πιο πιο αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Γι' αυτό το λόγο, με την εισηγήτρια την κυρία Μακοβέη και με την κυρία Αλφάνο, παρουσιάσαμε διάφορε τροπολογίε που προσθέτουν και ενισχύουν αυτήν την ε, πρώτη, το, πρώτο, το αρχικό κείμενο. Και έχουμε κάποιες θέσεις που παρουσιάζονται στο άρθρο 4, η τροπολογία 93. Έχουμε εισάγει την υπόθεση της διευρυμένης κατάστασης, εκεί όπου η δικαστική αρχή θεωρεί πως τα περιουσιακά στοιχεία του καταδικασμένου ατόμου είναι δυσανάλογα σε σχέση με την νόμιμη απασχόληση του συγκεκριμένου ατόμου και ότι αυτά τα αγαθά έχουν ε, αγοραστεί παρανόμως. Και όσον αφορά την κατάσχεση, την απουσία καταδίκης, έχουμε υποβάλει την τροπολογία 104 στο άρθρο 51 5.1α, ε, όπου προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών μελών να επιτρέψουν στι δικαστικέ αρχέ και τη απουσία ποινική ε, καταδίκη, να κατασχέσουν περιουσιακά στοιχεία ενό ατόμου που είναι κοινωνικά επικίνδυνη και που, α, που διεξάγει βίον ε, εγκληματικού τύπου. Όλα αυτά υπάρχουν στην Ιταλική νομοθεσία και είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν συγκεκριμένε διατάξει για να επιτραπεί η κατάσχεση τη απουσία καταδίκη σε συγκεκριμένε περιστάσει σε όλα τα κρατημέλη, καθώ και η αμοιβαία αναγνώριση αυτών των διαδικασιών. Και όσον αφορά τον προορισμό των κατησχεμένων ε, ε, περιουσιακών στοιχείων προβλέπεται ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να θετήσει τα απαραίτητα μέτρα με βάση τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται για να προβλέψει, να προλάβει την ε, απαλωτρίωση ε, του, των περιουσιακών αυτών Και μάλιστα δίνεται προτεραιότητα της χρήσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων για χρήσεις που παρεμποδίζουν την εγκληματικότητα ή για άλλες κοινωνικού τύπου χρήσεις, ούτως ώστε να επιτραπεί η αποτελεσματική δράση των, των Ευρωπαϊκών κρατών κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Στην Ιταλία έχουν φτιαχτεί ένα σωρό κοινωνικοί συνεταιρισμοί που εργάζονται και χρησιμοποιούν τα κατσχημένα περιουσιακά στοιχεία. Και όσον αφορά την κατάσχεση απέναντι σε τρίτους, τα ε, άρθρα 104, 125, άρθρο 4 ε, επιτρέπουν στις δικαστικές αρχές να κατασχέσουν ένα αγαθό ενός τρίτου. Μόνο όταν ο τρίτος αυτός ε, γνώριζε ή έπρεπε να γνώριζε πως αυτό το περιουσιακό στοιχείο ήταν το μέσο ή το πρόσοδο ενός εγκλήματος ή αν είχε επιλέξει δωρεάν μάλλον αν του είχε δοθεί δωρεάν ή σε πολύ χαμηλό υψηλότερη αξία από την πραγματική. Η τροπολογία 128 προτείνει στα κρατημέρη να υιοθετήσουν μέτρα που στόχο θα έχουν την ποινική δίωξη των όσων συμβάλλουν με εικονικό τρόπο, με αγαθά ή περιουσιακά στοιχεία που τα δίνουν σε τρίτους. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε κυρία Μποσελίνα. Ίσως η κυρία Λάτφορ θα θέλει να πάρει το λόγο. Um, Ευχαριστώ πρόεδρε, αλλά δεν είμαι σκιώδης της ομάδας. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Κατέθεσα κάποιες τροπολογίες. οι οποίες ε, εντάσσονται σε δύο κατηγορίες. Καταρχάς, ε, η μία κατηγορία έχει σκοπό να διευκρινίσει τα πράγματα γιατί κάποια κράτη μπορεί να είναι ποινικά τα θέματα αυτά αλλά κάποια κράτη τα εντάσσουν στο αστικό δίκαιο. Άρα κατέθεσα κάποιες τροπολογίες, όπως για παράδειγμα για μια εντελογική σκέψη που θα διευκρινίζει ότι η οδηγία που θα αφορά τέτοια μέσα δέσμευσης θα αφορά ποινικά ζητήματα και όχι αστικά ζητήματα προκειμένου αυτό να αναγνωριστεί, να διευκρινιστεί, όπως στην τροπολογία 91. Να διευκρινίσουμε ότι αυτή η διάταξη δεν ισχύει για κρατημέλη που έχουν αστικές διατάξεις για τέτοια δέσμευση και κατάσχεση προϊόντων για να διευκρινίσω ότι ενδεχόμενα μέτρα αστικού δικαίου, εθνικού αστικού δικαίου θα μπορούσαν να συνεχίσουν να υπάρχουν και να εφαρμόζονται. Και έτσι τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα είτε να ακολουθήσουν την αστική, την του αστικού δικαίου, είτε του ποινικού δικαίου χωρίς ε, καταδίκη. Οι άλλες τροπολογίες που κατέθεσα Ο σκοπό έχουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τις ε, σωστές ασφαλιστικές δικλίδες γιατί το Κοινοβούλιο έχει επεξεργαστεί διάφορα τέτοια μέτρα. Να μην επιδείξουμε λοιπόν έλλειψη συνοχής και συνεκτικότητας. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα τα οποία υπόκεινται τέτοια εντάλματα δεσμευσής θα πρέπει να απολαμβάνουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Εξού και η τροπολογία 138. Θα πρέπει το άτομο να έχει τη δυνατότητα να έχει, για παράδειγμα, νομική εκπροσώπηση. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την διάταξη αυτή. Επίσης, η 143, η τροπολογία μου 143, που αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα να αμφισβητηθεί αυτή, αυτό το ένταλμα, αυτή η εντολή ενώπιον ανεξάρτητης δικαστικής αρχής. Θεωρώ ότι αυτό συνάδει με τα υπόλοιπα μέτρα που έχουμε λάβει. Το B και το C. Ελπίζω να υποστηρίξει η Επιτροπή της τρόπολογίας αυτές ή κάτι παρόμοιο, εν πάση περιπτώσει. Τέλος, να αναφερθώ στην 147 τροπολογία που κατέθεσα που προτείνω να τροποποιηθεί το κείμενο γιατί δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα για τα μέτρα στο C άρα είναι μάλλον περίεργο να λέμε ότι θα πρέπει να εκπροσωπείται ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος των προϊόντων από δικηγόρο. Νομίζω ότι είναι περίεργο να λέμε ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να εκπροσωπείται από δικηγόρο. Μάλλον θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μπορεί, εάν θέλει, να εκπροσωπείται από δικηγόρο. Και στην 153 κυρία Μακοβέη προτείνω το δικαστήριο να εξετάζει κατά πόσον ένα άτομο θα υποστεί οικονομική καταστροφή σε περίπτωση δίμευσης των προϊόντων αυτών. Κατά πόσον δηλαδή ένα άτομο ενδεχομένως αν του στερηθεί η δυνατότητα να βγάζει το ψωμί του μπορεί τελικά να στραφεί στο έγκλημα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να δεχτείτε λοιπόν τις τροπολογίες αυτές. Κύριε Ταβάρις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Μακοβέ για τη συνεργασία που είχαμε και για τον επικοδομητικό διάλογο που είχαμε στη διάρκεια της εκπόνησης αυτού της έκθεσης και με τους άλλους σκιώδεις εισηγητές, με τους οποίοι, οι οποίοι μάλιστα πολύ ε, ε, είναι βαθύς γνώστες αυτής της ε, πραγματικότητας. Είναι πολύ σημαντική έκθεση αυτή. Όλοι μας καταλαβαίνουμε πως οι κοινότητες που άμεσα πλήττονται λόγω της ύπαρξης του οργανωμένου εγκλήματος πλήττονται άμεσα λόγω των εγκλημάτων αλλά και έμεσα λόγω της ε, ε, της ε, λανθασμένης χρήσης ή της κατάχρησης ε, πόρων που θα μπορούσαν ε, να χρησιμοποιηθούν για το κοινό καλό. Άρα λοιπόν πώς μπορούμε να κάνουμε νομικά τις κατασχέσεις, οι δημεύσεις και έπειτα τι να κάνουμε με τα κατασχεμένα προϊόντα, τα αγαθά, τα, τα στοιχεία. Η δική μου γενική εντύπωση είναι ότι συμφωνούμε όλοι όσον αφορά τους στόχους αυτής της οδηγίας δηλαδή εναρμόνιση της νομοθεσίας και δημιουργία μιας χρήσιμης βάσης ώστε να βλύνουμε και να αναχαιτήσουμε το έγκλημα. Η διχόνοια που μπορεί να έχουμε, οι διαφοράς που μπορεί να έχουμε, μπορεί να οφείλονται μόνο ε, σε κάποιες ε, διαφορετικές θέσεις ε, Όσον αφορά τη διαδικασία, η θέση της ομάδας μου είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο χώρο στο διάλογο και να βρούμε συνένεση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και την προσοχή που πρέπει να δώσουμε ώστε να μην φτιάξουμε μια νομοθεσία που κατά κάποιο τρόπο να ξεπερνά ή να υπερβαίνει κάποια νομικά όρια που είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας καταρχήν όσον αφορά το τεκμήριο αθωότητας το τεκμήριο αθωότητας που είναι η βάση, ο πυλώνας του κράτους δικαίου και θεωρώ πως υπάρχει τρόπος να, να φτιάξουμε και να υποδομήσουμε αυτή τη σχέση, αυτή την έκθεση με συγχωρείτε με τέτοιο τρόπο με βάση δηλαδή το τεκμήριο αθωότητας και μετά θα ήθελα να δω πιστεύω πως κάποιες τροπολογίες ιδιαίτερα η τροπολογία που ανέφερε πριν από λίγο η 104 που ανέφερε πριν από λίγο η κυρία Μπορσελίνο εγώ εν γέννη συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τη συνάδελφο Μπορσαλίνο. Μπορώ να πω και πολιτικά και ιδεολογικά για τα συγκεκριμένα θέματα, αλλά πιστεύω πως εκείνη η τροπολογία πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε τουλάχιστον να μπορούμε να εντοπίσουμε τα, τις να εντοπίσουμε υποκείμενα με βάση ένα στυλ ε, κοινωνικό, στυλ ζωής. Δεν νομίζω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάτι τέτοιο. Είναι πολύ ε, καθόριστο και αόριστο με τέτοιου είδους τροπολογίες. Δηλαδή όπως και με την 45 που λέει ότι η δυνατότητα δίμευσης μπορεί να υπάρχει ακόμα και τη απουσία καταδίκης. νομίζω πως είναι κάπως υπερβολικό. Πρέπει να έχουμε κάτι, ένα μήνυμο στοιχείο. Όπως τα είπα, είναι περισσότερο ε, ε, ένα θέμα μέσων, διαφορετικών μέσων για την επίτευξη του, ενός κοινού στόχου. Τώρα, για την κοινωνική χρήση των, των, των ε, δημευμένων περιουσιακών στοιχείων έχουμε μια τροπολογία που είναι η παριθμό 52 που λέει ότι οι ίδιοι πολίτες θα μπορούν να έχουν μια συμμετοχή συμμετοχή στην κοινωνική χρήση των κάτι σχήμα ε, ή δημευμένων περιουσιακών στοιχείων. Να είναι δηλαδή μια πτυχή πιο θετική, πιο δραστήρια αυτής της οδηγίας με κάποια στοιχεία της συμμετοχικής ε, δημοκρατίας. Αυτή είναι μια πρόταση που γίνεται με βάση που έκανε ε, το ίδρυμα που έκανε η το ελβετικό κράτος σε παράλληλα με το τραπεζικό του σύστημα για τη χρήση περιουσιακών στοιχείων που, κατα... τα οποία δημεύει και τα οποία συνήθως προέρχονται από δικτατορικά καθεστώτα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν Εάν έχουμε ένα ταμείο που αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία κατησχεμένα, δημευμένα, οι ίδιοι οι πολίτες να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με ένα, ας πούμε, μαζεύοντας υπογραφές ή, πάση περιπτώσει, να δίνεται προτεραιότητα στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από το οργανωμένο έγκλημα, ούτως ώστε οι πολίτες να βλέπουν, ναι, ότι το οργανωμένο έγκλημα πλήττει, ζημιώνει τις συγκεκριμένες κοινότητες, αλλά ναι, μπορούν αυτές οι ίδιες οι κοινότητες να συμμετέχουν κοινωνικά. Έχουμε και την 53, τροπολογία 53 διορθώνω και όχι 52 που είπα πριν. Και τέλος, να πω ότι στην περίπτωση που αυτές οι δημεύσεις ε, περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από έγκλημα ε, και πλήττουν κοινότητες εκτός της Ένωσης, γιατί συνήθω πρόκειται για κοινότητε εντός. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν μήπω τα, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να ωφελήσουν ε, τι κοινότητε που έχουν ε, ζημιωθεί με αναπτυξιακά προγράμματα, όταν πρόκειται δηλαδή για εξοκοινωτικές ε, κοινότητε που έχουν ζημιωθεί. Σα ευχαριστώ πολύ και στην διατύπωση των συμβαστικών τροπολογιών μπορούμε να βρούμε συνένεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέρκοπ. Ευχαριστώ, θα είμαι. Είστε σκιώδη γιατί θυμίζω. Ναι, κύριε Σκύρου, θα είμαι πολύ σύντομο, δύο σημεία, πολύ γρήγορα. Το πρώτο είναι ότι για το θέμα αυτό το σημαντικότερο, τη δική μου τουλάχιστον ε, οπτική γωνία, είναι ότι υπάρχει ή να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση για τα εντάλματα δίμευση κατάσχεση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ανά την Ευρώπη για την επιβόληση της νομοθεσία. Το δεύτερο σχόλιο αφορά το ότι ενώ από την νομική υπηρεσία καθίσατε σαφές ότι αν υπάρχει ε, σχέση με την εγκληματική δραστηριότητα, στηρίζω τη δραστηριότητα, την ανθρωπολογία 91, πάλι συμφωνώ με αυτά που λέει η κυρία Λάτφορντ. Θεωρώ ότι εκεί όπου υπάρχουν συστήματα και το αστικό δίκαιο είναι αυτό το οποίο είναι ο φορέας, ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να παρέμβουμε στις δραστηριότητες τους. Ε, αυτό είναι σημαντικό και νομίζω ότι θα ήταν και πάρα πολύ περίπλοκο να επιβάλλουμε σε χώρες να δώσουν ε, ποινικέ εξουσίες ενώ υπάρχουν ε, μέσω της αστικής διαδικασίας, των διαδικασιών αστικού δικαίου ή εάν δεν, θεωρούν, δεν θεωρούνται ότι πληρούν τέτοια μέτρα της δραματεύσεις της νομικής υπηρεσίας. Αμοιβαία αναγνώριση λοιπόν είναι το βασικό για μένα. Ευχαριστώ. Και τροπολογία 91. Vielen Dank. Ähm, Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία και να πω ότι μπορεί να ε, έχει μεγάλη προθυμία, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουμε και ε, μια προσεκτική στάση σε περίπτωση κατάσχεσης χωρίς ε, ε, καταδίκη. Είναι τόσο ευαίσθητο το θέμα αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ για να μην ε, απαρνηθούμε βασικές αρχές του ποινικού δικαίου όπως το δεκμήριο αθαότητας, το δικαίωμα, τα περιουσιακά στοιχεία, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Τέτοια λοιπόν κατάσχεση χωρίς καταδίκη θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή. Γιατί κάθε τι άλλο θα ανέτρεπε το τεκμήριο αθωότητας. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να τονίσω την τροπολογία 36 της Σάρα Λάτφορντ να αναφερθεί ότι διευκρινίζουμε ότι πρόκειται για ποινικά ζητήματα και όχι για αστικά ζητήματα. Επίσης, διαπιστώνω ότι πολλές τροπολογίες εντοπίζουν τα ίδια προβλήματα από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Σημαντικό είναι, για παράδειγμα, η τροπολογία 56 σε ό,τι αφορά τις σχετικές ρήτρες σε ό,τι αφορά την αναγκαστική κατάσχεση. Αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει μεγάλο αντίκτυπο. Άρα χρειάζεται η ρήτρα αυτή, ιδιαίτερα όταν τα μέτρα επιβαρύνουν δυσανάλογα. Είτε τον ε, κατηγορούμενο είτε τα θύματα. Ένα δεύτερο θέμα τα άρθρα 4 και 5 για την ε, εκτενή κατάσχεση χωρίς καταδίκη. Θεωρώ ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Θεωρώ ότι στην παρούσα φάση το άρθρο αυτό δεν διατυπώνεται με επαρκή ακρίβεια και η κατάσχεση και η κατάσχεση χωρίς ε, καταδίκη θα πρέπει να τηρούν κάποια ελάχιστα ποινικά πρότυπα θεωρώ ότι χρειάζεται πιο καλή διατύπωση για να διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται αυτή η κατάσχεση χωρίς καταδίκη εφόσον το δικαστήριο έχει πιστεί βάσει συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων. Σε περίπτωση που μιλάμε για κατάσχεση χωρίς καταδίκη να θεωρεί το δικαστήριο ότι θα ακολουθούσε καταδίκη σε περίπτωση εκδίκασης. Στο άρθρο 7, ένα σημείο στο οποίο έχω θέσει δύο για την παραγραφό 1 και 2 που συνοψίζονται προκειμένου να γίνουν πιο συγκεκριμένες. Τέλος, πολύ αμφισβητούν την χρήση των ε, ε, αξιών περιουσιακών στοιχείων. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν εντάσσεται σε καμία περίπτωση στον τομέα εφαρμογή της οδηγίας αυτή. Το θέμα είναι να βρούμε ελάχιστα πρότυπα για την ε, κατάσχεση αυτή. Αλλά τώρα το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα ποσά αυτά θεωρώ ότι δεν ταιριάζει στην οδηγία αυτή. Στη Γερμανία τα ποσά αυτά θα χρησιμοποιούνταν για προς των θυμάτων, για παράδειγμα. Αλλά νομίζω ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να κληθεί να αποφασίσει τι θα κάνει με τα ποσά αυτά. Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών προϋπολογισμών δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί σε τέτοια συνάρτηση. και όταν μάλιστα πρόκειται για τέτοια παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του εκάστοτε ατόμου. Ευχαριστώ κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εν συντομία, για να μην επαναλάβω άλλωστε όσα έχουν ήδη υποθεί. Αδιαφυσβήτητα πρόεδρε. Το νέο είδος ε, διασυνοριακού εγκλήματος χρειάζεται και τα κατάλληλα νομικά μέτρα και μέσα για να το αντιμετωπίσουμε. Όλοι συμφωνούμε από αυτού. Εκ παραλίλου θα πρέπει να επιτύξουμε μεγάλη προσοχή στη διαδικασία αυτή. δάλος διακυβεύεται ό,τι έχουμε πετύχει στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δεκαετία του 1950. Και μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε κανόνες σαφείς όμως. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες και οι ίδιοι δικαστέ. Και αυτό ισχύει για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή ζήτησε από την υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων να γνωμοδοτήσει. Και νομίζω ότι πολλές από τις τροπολογίες που έχουν κατατηθεί συνάδουν με τα πορίσματα της υπηρεσίας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα σε ό,τι αφορά την εκδίκαση αποτελούν δικαιώματα θεμελιώδη. Όταν μιλάμε για το τεκμήριο αθωότητας, ε, το δικαίωμα δίκαιης δίκης, εκπροσώπησης από δικηγόρο και ούτω καθεξής. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η αναλογικότητα ασφαλώς των μέτρων. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όποτε χρησιμοποιείτε το μέτρο αυτό, χρησιμοποιείτε λόγω πολύ βασικών αδικημάτων. Γιατί αν κάνουμε μία εξαίρεση σήμερα και άλλη μία σε τρία χρόνια, πού θα καταλήξουμε σε 20-30 χρόνια. Σε έναν πολύ διαφορετικό κόσμο. Αυτό δεν νομίζω ότι το επιθυμούμε. Επίσης, εγώ προσωπικά κατέθεσα μία σειρά τροπολογιών συνάδουν λίγο πολύ με τις άλλες τροπολογίες των συναδέλφων. Νομίζω ότι θα διευκολύνει το έργο μας για το μέλλον. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για τις προσπάθειες για συμβαστικές τροπολογίες. Θεωρώ ότι είναι ευκταίο τελικά η έκθεση να αποτυπώνει τις απόψεις όλων των πολιτικών ομάδων προκειμένου να μην καταστεί ιδεολογικό το ζήτημα. Γιατί όπως σας είπα είναι σημαντικό να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα αλλά και να προασπίσουμε τα δικαιώματά μας. Thank you. Ευχαριστώ κυρία Ματιέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κείμενο που έχουμε αναχείρας. Το είχαμε ζητήσει και ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της ε, συγκρότησης και της Επιτροπής ΚΡΙΜ. Κάτι που είχε ζητήσει η Επιτροπή ΛΥΠΕ και πέρυσι είχε ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Ορισμένοι συνάδελφοι παρόντες, Μακοβέη, Μπορσαλίνο, δεν ξέρω αν είναι κάποιος εκεί, Ταβάρες, ναι, και τα λοιπά που είναι μέλη και της Επιτροπής ε, ΚΡΙΜ όπως και εγώ. Πρέπει να σας πω ότι καλό θα ήταν να έρθετε και άλλοι στην Επιτροπή Κρίμου. Γιατί νομίζω ότι τότε θα θετούσατε μια εντελώ διαφορετική προσέγγιση. Η κυρία Προσολίνο και η κυρία Σμακοβέ βλέπουμε ότι δεν έχουν τις ίδιε απόψεις ε, με άλλους συναδέλφου. Ίσως ε, εμείς θα θέλαμε να είναι λίγο πιο αυστηρό το κείμενο. Βέβαια πάντοτε θέλουμε να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθότητας, αλλά εγώ προσωπικά χωρίς να έχω κάνει καμία περιδάσκηση σε, σε κάποιο δικαστήριο παρά στη Γαλλία. Τουλάχιστον ξέρω ότι έχω την εντύπωση ότι οι δικαστές εργάζονται διαφορετικά, αλλά σέβονται και το, την αρχή του τεκμηρίου αθότητας. Η γαλλική δικαιοσύνη λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Όταν βλέπουμε λοιπόν τη δραστηριότητα της μαφίας στην Ευρώπη και όχι μόνο, νομίζω θα μπορούσαμε πραγματικά να κάνουμε λίγο πιο αυστηρό το κείμενο, να διευρύνουμε την δίμευση και την κατάκτηση mm. των περιουσιακών στοιχείων, αλλά και το πάγωμά τους. Αυτό θα διευκόλυνε την εκτεταμένη δίμευση, γιατί όταν ακούμε, δεν ξέρω, εδώ και εξι μήνες, 6-7 μήνες το επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό στην Επιτροπή Κρίμ και έχουμε κρουαστεί εγκληματολόγους, εμπειρογνώμες από την Europol, από την Όλαφ κτλ. Βλέποντας λοιπόν τη δραστηριότητα αυτής της μαφίας, της διακρατικής μαφίας, βλέπουμε ότι πραγματικά υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ένας από τους τελευταίους εγκληματολόγους που είχε έρθει σε μια κρόαση έλεγε ότι πιο πολλού νεκρούς δημιουργεί πλέον στην Ευρώπη η οργανωμένη μαφία, το οργανωμένο κλίμα και όχι τόσο η τρομοκρατία. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η δραστηριότητα και η συμπεριφορά της μαφίας. Για τα χρήματα τα κάνουν όλα αυτά. Δεν πρέπει να το ε, ξεχνάμε αυτό και για την αγορά ε, ακινήτων και, άλλων, και, και άλλων αγαθών. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε τη δράση της Μαφία πέραν των όσων κάνουν. Σίγουρα πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματα ε, των προσώπων και τα το τεκμήριο της αθωότητας. Εδώ όμως έχουμε ένα κείμενο για να βοηθήσει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της μαφίας. αλλά εγώ από το κείμενο και από τις συζητήσεις βλέπω ότι πιο πολύ καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και κάπως προστατεύουμε και τη μαφία. Ενώ έχουμε τη δυνατότητα να αγωνιστούμε και να κάνουμε κάτι. Λίγο με απογοητεύουν όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι όλοι μας ε, αγωνιζόμαστε κατά της μαφίας, ε, είμαστε πολύ προσιλωμένοι σε αυτό το στόχο. Μας υποβάλλει ένα κείμενο η Κομισιόν, έχουμε τη δυνατότητα να ε, έχουμε στα χέρια μας ένα ενδιαφέρον νομοθετικό εργαλείο και παρόλα αυτά τελικά μένουμε στη μέση είμαι λίγο απογοητευμένη. Αν δεν έχουμε το θάρρος να προχωρήσουμε, δεν ξέρω εγώ, ε, θα είμαι ε, απογοητευμένη τελικά. Θα ήθελα, νομίζω και η κυρία Μακοβέκη και η κυρία Μπροσαλίνου θα το ήθελε, να προχωρήσουμε και να καταπολεμήσουμε και με νομοθετικό πλέον ε, τρόπο τη μαφία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Μπόκουρτ. Κυρία Μπόκουρτ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Μακοβέη, για τη σημαντική της δουλειά, για το σημαντικό αυτό θέμα και εγώ κατέθεσα τραπολογίες να συμφωνήσω με τη συνάδελφο Ματιέ ότι προπαντός σημαντικό είναι να έχουμε ένα αποτελεσματικό μέσο στα χέρια μας. Οι τροπολογίες μου, όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι, σκοπό έχουν να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα, που, τα προσωπικά στοιχεία τα οποία δημεύονται. Ακολουθούν τη σωστή διαδικασία. Το είχαμε τονίσει αυτό και σε ό,τι αφορά την εμπορία των ε, ατόμων. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε και εδώ. Και τέλος. Αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί και το θέλουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των αρχών της εφορίας, της αστυνομίας, του δικαστικού σώματος για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί όντω. Ελπίζω λοιπόν οι συνάδελφοι να υποστηρίξουν τι τροπολογίε αυτέ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπορσελίνο θέλει να επανέλθει. Σύντομα όμω, πριν να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Ε, δεν θα σχολιάσω τις ε, παρεμβάσεις ε, των συναδέλφων ήταν όλες πολύ ενδιαφέρουσες και όσον αφορά εμένα δεν μπορώ να αμφισβητήσω καθόλου τα θεμελιώδη δικαιώματα εννοείται όλων όμως όχι μόνο των ε, ε, κατηγορούμενων εγκληματιών αλλά και για των ανθρώπων και τη κοινωνίας πέρα από τα θύματα τα ίδια και να κάνω μια άλλη παρατηρήση η ημερομηνία της ψηφοφορίας έχει οριστεί για τις 31 Ιουνίου όμως η 31 Ιανουαρίου η ομάδα των σοσιαλιστών συνεδριάζει στην Τεργέστη. Άρα δεν θα μπορούμε να έρθουμε να ψηφίσουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή ξαφνικά να έρθουμε πίσω στο κοινοβούλιο. Τι θα κάνουμε. Όλη η ομάδα των σοσιαλιστών συνεδριάζει στην Τεργέστη. Sì, proprio vero. <laughs> vero. <laughs> ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Ναι, πριν να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, μάλλον, α, ο κύριος Ταβάρες θέλει ακόμα το λόγο. Ναι, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. για το μέσο. Φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, αλλά έχω μια διαφωνία με τον Axel Voss για το στόχο και νομίζω πως αυτή η διαφωνία μπορεί να είναι προπαραγωγική. Αν θέλει κανείς να κάνει περίπλοκη και δραστήρια καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο θα πρέπει κανείς να σκεφτεί την κοινωνική χρήση αυτών των ε, περιουσιακών στοιχείων ως μέσο καταπολέμησης του εγκλήματος. Θα πρέπει να είναι τμήμα λοιπόν όλα αυτά. Ε, δηλαδή, η, ε, ο αντίκτυπος του οργανωμένου εγκλήματος είναι τόσο βαθύς, ε, κοινωνικά και ιστορικά, και το είδος λοιπόν του αγώνα που, θες να, που θα πρέπει να κάνει κανείς δεν είναι μόνο νομικού και αστυνομικού τύπου, επιβολή νόμου, αλλά θέλεις και να αλλάξεις αυτόν τον τρόπο ζωής και ένας τρόπος είναι να ε, τη, η νόμιμη χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων να αποδειχτεί πως είναι καλύτερη από αυτή που γίνεται από το οργανωμένο έγκλημα. Και ένα ακόμα σχόλιο, ότι φυσικά αυτό που λέμε όταν ε, μιλάμε για δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου να ε, αποτελείται αυτό από ένα κομμάτι των κατσχημένων ε, περιουσιακών στοιχείων. Δεν μπορούμε να έχουμε διπλά σταθμά εδώ. Να, δεν μπορούμε να ζητάμε από την Ένωση να ενεργεί και να νομοθετεί, να προβαίνει σε αστυνομική και δικαστική συνεργασία και μετά το να υπάρχει ένα σχετικό Ευρωπαϊκό Ταμείο να είναι ταμπού και όλα τα κατασκευμένα αγαθά που κατάσχονται με ευρωπαϊκή δράση, ευρωπαϊκή συνεργασία και ευρωπαϊκή νομοθεσία να επιστρέφουν στα κράτη-μέλη μόνο. Εντάξει, ένα κομμάτι να πάει σε ένα ευρωπαϊκό τομείο, ώστε να πούμε στους, ευρωπαϊκούς, στους ευρωπαίους πολίτες ότι η κοινωνική χρήση ανήκει στην κοινότητα που είναι τοπική, εθνική και διεθνής ε, και θα πρέπει να είναι κομμάτι αυτό του προβληματισμού μας. Ευχαριστώ. Είναι εδώ ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μπορείτε να μας ε, παρουσιάσετε λίγο το πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη χρονική στιγμή. Σύντομα όμως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους σκιώδη εισηγητή, αλλά και όλα τα άλλα μέλη τη Επιτροπής ΛΥΠΕ για τι τροπολογίε που κατέθεσαν και για την οικοδομητική του συμβολή. Από ό,τι προκύπτει από τη συζήτηση αυτή είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Η Κομισιόν έκανε ό,τι μπορούσε για να υποβάλει μια ισορροπημένη πρόταση ώστε να καλυφθούν οι, καλυφθεί τεράστιο φάσμα λύσεων που υπάρχουν στα κρατημέλη σε ό,τι αφορά τη δίμευση περιουσιακών στοιχείων. Εμείς προσπαθήσαμε να προτείνουμε ένα μέσο το οποίο θα αποτελεί προστιθέμενη αξία. Και το θέμα είναι να πετύχουμε το βασικό, το βασικό μας στόχο που είναι το οργανωμένο έγκλημα. Και έχει, ξέρουμε, έντονη ε, διασυνοριακή διάσταση το οργανωμένο έγκλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα ε, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα κάνω κάποια σχόλια, όχι όμως ε, αποσκοπώντας να καλύψω τα πάντα. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 66, 67 μάλλον και 68, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι η διήμευση κατάσχεση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για τα άμεσα έσοδα εγκληματικών δραστηριοτήτων, αλλά να τηρούνται ε, οι διατάξει των διεθνών συμβάσεων. Άρα θα πρέπει να μπορεί να αφορά και περιουσιακά στοιχεία τα οποία επενδύθηκαν σε άλλε ε, μη άμεσα σχετιζόμενα ε, δραστηριότητε και άρα αποτελούν και αυτά παράνομη περιουσία. Είμαστε στο πλαίσιο της νομικής βάσης όπου ορίζεται η δίμεση ως ποινή. Όμως, ταυτόχρονα, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η κατάσχεση, αυτή η δίμευση θα μπορεί να καλύπτεται και να αφορά μάλλον και άλλα, όχι ε, από προερχόμενα επαγγελματικές δραστηριότητε ε, έσοδα. Και τι θα πρέπει να γίνει σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να δημευθούν τα στοιχεία τα οποία αποτελούν παράνομους προσόδους. Είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Επίσης, θέλουμε να τονίσουμε ότι η μη καταδίκη, η τροπολογία 90 αλλά και η τροπολογία 4 της ηγετρίας που προτείνει να έχουμε κατασχέσεις μη βασιζόμενες σε καταδικαστικές αποφάσεις ή απουσία κάποιας δίκης, για παράδειγμα. Εγώ ε, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε ειδικέ περιπτώσεις όταν δεν θα μπορεί να υπάρξει ποινική δίωξη. Γιατί αλλιώς ε, νομίζω ότι υπερβαίνουμε την εντολή που μας ε, έχει δοθεί μέσω των συνθήκων. Επίση έχουμε κάποιε ανησυχίε για τις τροπολογίες που ζητούν να παρασκευθεί πλήρε ε, αποδεικτικό υλικό. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να διακινδυνεύσει την ίδια την αρχή της εκτεταμένη δίμευσης που στα περισσότερα κράτη-μέλη ισχύει και έχει ενταχθεί πλέον στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά όχι με απόλυτα σαφή τρόπο ακόμη. Μια πάρα πολύ σημαντική για εμάς διάταξη και είναι και ένα κρίσιμο τεστ, αν θέλετε, για τη διαδικασία ε, αυτή της ε, μη βασιζόμενης δίκη δίμευση. Δεν θα θέλαμε να εφαρμόζεται, παραδείγματος χάρη αυτή η δυνατότητα για περιπτώσεις όπου ο εναγόμενος ε, έχει αποβιώσει, για παράδειγμα. Θα ήταν αυτό επικίνδυνο διότι θα μπορούσε η κοινωνία να μην αποφεληθεί από τεράστια ε, ποσά που αποτελούν προϊόν παράνομη δραστηριότητα και δεν μπορεί να τα εκμεταλλευτεί. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες ε, περαιτέρω, αλλά να, να σας πω ότι ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο με τα ένδικα μέσα, με τα εχέγγυα που έχει αυτό το κείμενο, θα τα διατηρήσει. Για πρώτη φορά έχουμε μια πολύ σημαντική οδηγία στο ποινικό δίκαιο. Που βέβαια πρέπει να ε, συμπληρωθεί γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα με τα απαραίτητα εχέγγυα. Σας ευχαριστώ πάντως που μου δώσατε το λόγο και προσβλέπουμε και εμείς στη συνέχεια των ε, διαπραγματεύσεων αλλά και βασιζόμαστε στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου γιατί ξέρετε αν υπάρξει αυτή η συνθήκη θα αλλάξει επιτόπου την όλη κατάσταση. Πρόεδρος, η Ιρλανδική Προεδρία θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ξέρετε ότι το Συμβούλιο έχει καταλήξει σε μια γενική προσέγγιση για το θέμα αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την Ιρλανδική Προεδρία και αφορά ιδιαίτερα τον Υπουργό Δικαιοσύνης ε, Ισότητας που θα έρθει στην Επιτροπή σας τις επόμενες εβδομάδες. Ελπίζουμε να σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Κοινοβούλιο και χαιρόμαστε που η συγγήτρια και οι σκιώδες εισηγητές ε, έχουν σημειώσει πρόοδο. Στην πρώιμη αυτή φάση θα ήθελα να σας πω ότι ασφαλώς και δεσμευόμαστε να προχωρήσει το θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε και εμείς, ε, λέει ο Πρόεδρος και τώρα η κυρία Μακοβέη έχει και πάλι το λόγο. Βλέπω ότι έχετε σημειώσει τα θέματα τα οποία ε, ανέφερε κυρία Μπορσελίνο. Πρόκειται για μια προγραμματισμένη συνάντηση των σοσιαλιστών σε ό,τι αφορά την μετάβαση στην Τριέστη 30 και 31 του μηνός. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε για να τους διευκολύνουμε, γιατί είναι εξίσου σημαντική αυτή η συνάντηση, όπως οι συναντήσεις όλων των ομάδων αλλά τα μέλη της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ θα πρέπει να μεταβούν στον Τριέστη. Αν λοιπόν κάτι μπορείτε να κάνετε, να μας διευκολύνετε κυρία Μακοβέη, ευχαριστώ λέει κυρία Μακοβέη. Μία λύση θα ήταν να έρθουμε όλοι μαζί στην Τριέστη για να ψηφίσουμε. Ναι, ναι, ναι, κοιτάξτε. Θα το συζητήσω με τη γραμματεία για να βρούμε μια κατάλληλη ημερομηνία που να βολεύει όλους τους συναδέλφους. Κάποια σχόλια, επιτρέψτε μου. για μένα, την κυρία Μπορσελίνο και την κυρία Αλφάνο. Το πιο σημαντικό εδώ στην οδηγία είναι η κατάσχεση χωρίς καταδίκη, η εκτεταμένη κατάσχεση και η κατάσχεση τριών μερών. Γιατί μετά από καταδίκη η κατάσχεση που περιορίζεται στο αντικείμενο εγκληματικής καταδίκης για το οποίο υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι αποτελεσματικοί. Δεν αρκεί. Και τελικά τα χρήματα μένουν στους κόλπους των εγκληματικών αυτών οργανώσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Και αυτό συνάδει με αυτά που είπε και η κυρία Ματιό και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Επίσης, να θέσω και το προσωπικό μου στοιχείο. Τα καλύτερα συστήματα θεωρώ είναι στον Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία σήμερα, όπου η κατάσχεση γίνεται μέσω αστικής ε, διαδικασίας. Μπορούμε να πούμε ότι η πράξη είναι ποινικό, ποινικής φύσεως, άρα τελικά απευθύνεται κανείς στα αστικά δικαστήρια. Είναι μεγάλη η γκάμα της νομοθεσίας που ισχύει σε κάθε κρατός μέλος. Αυτό το είδαμε και σήμερα, μίλησε το κάθε μέλος της Επιτροπής μας. Νομίζω ότι τελικά θα πρέπει και καλούμαστε να βρούμε μία λύση για όλη την Ένωση. Δεν είμαστε εδώ προκειμένου να τροποποιήσουμε το κάθε νομικό σύστημα, αλλά για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Και ναι, τελικά κάποια κρατημέλη θα κληθούν να τροποποιήσουν την νομοθεσία τους. Όντως, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές δικλείδες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάθε τέτοια κατάσχεση θα πρέπει να γίνεται από δικαστήριο. Ας το συζητήσουμε, αλλά έχει αποφασιστεί εξ αρχής αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Να πω επίσης πληροφοριακά για τους συναδέλφους ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκε σε διάφορες περιπτώσεις ότι η κατάσχεση βασιαστικών ε, μέτρων συνάδει με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Θα το συζητήσουμε λοιπόν. Θα συζητήσουμε τις προτινόμενες συμβαστικέ προτάσεις, αλλά θα ήθελα εκ νέου να τονίσω ότι η πρόθεσή μου είναι να προχωρήσουμε με ένα δυνατό κείμενο σε ό,τι αφορά την κατάσχεση χωρίς καταδίκη, την εκτεταμένη κατάσχεση και την κατάσχεση από τρίτα μέρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος, που συνοψίσατε τα συμπεράσματά σας. Ασφαλώς και για τη συνεργασία σας και σε ό,τι αφορά την ημερομηνία ψηφοφορία. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρο. Έτσι ολοκληρώνουμε το τελευταίο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Επόμενη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ στις 21 Ιανουαρίου, 3 η ώρα το μεσημέρι, 21 και 22 Ιανουαρίου θα συζητηθούν εκ νέου τα ζητήματα αυτά. Ευχαριστώ.